well, good morning, everybody. Could I, um, could I invite you to take your places? Καλημέρα, παρακαλώ καθίστε. Έχουμε δύο από τους εισηγητές μας εδώ. Δεν ξέρω που είναι ο κ. Μπουσό. Η τη φαντάζομαι. Uh, so, very warm welcome to everybody to our committee this morning. Καλώς ήρθατε όλοι στην σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε μπροστά μας μια πλήρη, ολόκληρη μέρα εργασίας. Το πρωί θα εξετάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό κείμενο της, ε, του νόμου για την ενιαία πράξη. Όπως πολύ γνωρίζετε η Επιτροπή μας αποφάσισε λόγω του, της πολύ σημαντικής ε, πρωτοβουλίας που αντιπροσωπεύει αυτό το νομοθετικό κείμενο και στο οποίο εμπλέκονται πολλές επιτροπές να γίνουν τρεις εκθέσεις που, θα καλύπτει κάθε μία το κάθε κεφάλαιο. Έχουμε την κυρία Κανιέρη, τον κύριο Ντεκάμπος, ελπίζω να έρθει ο κύριος Μπουσόη και οι τρεις ηγητές μας θα είναι παρόντες. Συνεργάστηκαν και στενά μεταξύ τους, διότι θα είναι ένα συντονισμένο έργο όλη της επιτροπή, θα, θα συναντώνται οι συντονιστές με τους εισηγητές, τόσο ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο τελικά. Επίσης, καλέσαμε εκπροσώπους στην συνάντηση από άλλες επιτροπές, ιδίω τι επιτροπέ, που έδειξαν ενδιαφέρον και καλωσορίζω τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, τον κύριο Σίμψον, πολύ καλό φίλο μου μεταξύ άλλων, και θα του δώσει την ευκαιρία να μιλήσει εξ ονόματο τη Επιτροπής του ε, για να συμβάλλουν και αυτές στο έργο μας. Κάποια τυπικά στοιχεία. Υποθέτω ότι εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη, νομίζω. Δεύτερον, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η συνάντηση αυτή είναι σε web stream και θα σας ζητούσα λόγω του webstream να, να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο που είναι στα αριστερά σας αν ε, δεν το έχετε ακριβώς μπροστά σας λόγω των, ε, της οπτικής γωνίας της κάμερας. Θα το ελέγξουμε πάντως αυτό. Καλωσορίζω όλους όσοι μας παρακολουθούν από το ίντερνετ και στα ντοσιέ σα έχετε δύο ομάδες πρακτικών από προηγούμενες συναντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο των πρακτικών, αύριο το μεσημέρι θα εγκριθούν. Αυτή είναι η σημερινή διαδικασία. Η κυρία Στάιλερ θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κοιτάζω την ημερήσια διάταξη Πιστεύετε ότι έχουμε αρκετό χρόνο για τις πληροφορίες σήμερα το απόγευμα, γιατί έχουμε την οδηγία για τα δικαιώματα καταναλωτή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο από ό,τι φαίνεται στην ημερήσια διαταξία τις ψηφοφορίες. Δεν το ξανασκέφτεστε. Το είδαμε όταν ε, κοιτάζαμε τα τις ψηφοφορία. Οι σκιώδεις συγκεκριτές έκαναν καλή δουλειά στις συμβαστικές τοπολογίες και πιστεύω ότι είναι ελέγξιμος ο αριθμός των τροπολογιών μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες μετά τις 6.30 αν χρειαστεί χωρίς διερμηνία. σε αν χρειαστεί κάτι τέτοιο θα το αποφασίσουν οι, συγητές, οι συντονιστές. Συγγνώμη. Μπορεί νομίζω να γίνει, να συνεχιστεί η ψηφοφορία έστω και χωρίς ε, διερμηνία, αλλά... Ελπίζω και ευελπιστώ ότι οι συντονιστές θα προωθήσουν γρήγορα την έκβαση της συζήτησης. Να είστε πάντως όλοι εδώ με τις κάρτες σας και να προσέχετε και εμένα και τους συντονιστές σας για τα, για τα μηνύματα που σας στέλνουν για να προχωρήσουμε γρήγορα. Ε, θα ήθελα με την ευκαιρία να υπενθυμίσω σε όλους να είστε στην ώρα σας το απόγευμα. Επίσης έχουμε ε, τρία τέταρτα συνάντηση με τον Επίτροπο Καινοτομίας κ. Κουίν στο ξεκίνημα της απογευματινής συνάντησης και τώρα και σε αυτό να είστε επακριβείς διότι πραγματικά η κυρία Κουίν ε, μας τίμησε με την επίσκεψη στην Επιτροπή ιδιαίτερα για τα θέματα των δημοσίων ε, συμβάσεων και την χρήση της καινοτομία της δημοσίες συμβάσεις που ήταν κάτι που ζητούσαμε στην Επιτροπή και είναι εξαιρετικά χρήσιμο ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει και μια πρόταση της Επιτροπής υπομορφή πράσινης βίβλου που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα οι συντονιστές συμφώνησαν να ζητήσουμε να ξεκινήσουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την πρόταση αυτή εξ αρχής. Εφόσον εγκριθεί η, κυρία, η έκθεση της ε, ε, κυρία Σάλντε Μόζε σήμερα το απόγευμα, θα ζητήσω από την Επιτροπή να ξεκινήσουμε άμεσα για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτές είναι οι αναγγελίες του Πρόεδρου. Τι προτείνω. Πρώτον, να πάμε κατευθείαν στη συζήτηση για τις εκθέσεις. Θα δώσω το λόγο στους τρεις εισηγητές για να παρουσιάσουν το πλαίσιο και τα θέματα των εκθέσεών τους. Κατόπιν θα ξεκινήσουμε την συζήτηση και αν συμφωνεί ο κύριος Σίμψον θα του δώσω και την ευκαιρία να, μπει, να μιλήσει πρώτος γιατί φαντάζομαι ότι έχει και άλλες δουλειές. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος επιτροπής. Θα του δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές για οποιαδήποτε από τις τρεις εκθέσεις και στους σκιώδεις άλλων επιτροπών που είναι παρόντες. Και μετά θα παρέμβουν και οι ίδιοι οι θα το δούμε και στη μέση πώς προχωράει. Θα υπάρχει αρκετό χρόνος πάντως. Εάν συμφωνείτε, θα ζητήσω από την κυρία Σάντρα Καλνιέτε να ξεκινήσει τη συζήτηση. Κυρία Καλνιέτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε το σχέδιο για την, ε, το τμήμα της έκθεσης για τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους, ιδίω τους και τους για τις ιδέες που πρότειναν. Θα ήθελα να σας πω ότι έλαβα σχόλια από όλες σχεδόν τις πολιτικές ομάδες, ιδίω ε, θέλω να αναφέρω την βοήθεια της γραμματείας και του κύριο Κούγκλα καθώς και της ε, συμβούλου του ΕΛΚ, της κυρίας Τερέζα Ντεπίντου. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις όλων λόγω του ότι ωστόσο το σχέδιο δεν έπρεπε να ξεπεράσει τους 6.000 χαρακτήρες, ήταν περιορισμένο δηλαδή, δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα σχόλια. Είμαι βέβαιη ωστόσο ότι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την έκθεση με τις τροπολογίες σας. Κάποια από τα θέματα που δεν ταιριάζουν στο κύριο κείμενο της έκθεσης αντιμετωπίστηκαν στα, στην, ε, αιτιολογική έκθεση, ιδίω το Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά. Και προτείνω, προτίθεμαι να υποβάλω δική μου τοπολογία για να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο η πρώτη αυτή στην έκθεση. Να πω δύο λόγια για τη δομή. Πρώτον, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσόη και τον κύριο Ντεκάμπος για την υποδειγματική συνεργασία τους και το πνεύμα βοήθειας που είχαμε μεταξύ μας στις διαβουλεύσεις και οι τρεις συμφωνήσαμε να προτείνουμε μια παρόμοια δομή και για τις τρεις εκθέσεις ε, που περιλαμβάνουν την εισαγωγή σαν πρώτο τμήμα, ένα δεύτερο τμήμα με την αξιολόγηση των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή με την νομοθεσία για την ενιαία, για την αγορά στο τμήμα διακυβέρνησης και εταιρικών σχέσεων και να κλείσω την έκθεση με ένα τρίτο τμήμα που αφορά τις βασικές προτεραιότητες δράσεων που προτείνουν οι εισηγητές, ο κάθε εισηγητής ξεχωριστά. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, ε, για να αποτελέσουν πραγματικές προτεραιότητες θα ήταν σκόπιμο να περιοριστούν σε πέντε το πολύ 7 ανά έκθεση. Τώρα, για την διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση κάποια λόγια. Υποστηρίζουμε τις περισσότερες προτάσεις της Επιτροπής και περαιτέρω ενισχύουμε ορισμένες από αυτές. Ποιε είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις. 1. Ισχυρότερη πολιτική ηγεσία. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να αυξηθεί το πολιτικό προφίλ και η δημόσια επίγνωση της σημασίας της ενιαία αγορά. Γι' αυτό υπογραμμίζω την ανάγκη να υπάρξει παρότρινση και ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, εφαρμογή της Στρατηγικής Ένωση 2020 και επανα... επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς. Και οι τρεις αυτές τις προτεραιότητες είναι εξίσου σημαντικές για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε από τα κράτη-μέλη να, να, δεχθούν και να γίνουν κύριοι της νέας όθεσης της ενιαίας αγοράς. Προτείνουμε ο πρόεδρος του Συμβουλίου να αναλάβει την εντολή να συντονίζει και να εποπτεύει την νέα εκκίνηση της ενίας αγοράς και ζητούμε κάθε ανεξάρτητη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφιερώνεται στην αξιολόγηση της παρούσης καταστάσεως της ενίας αγοράς. Επίσης, υπογραμμίζουμε τον ενισχυμένο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην διαδικασία έγκρισης νομοθεσίας της Ένωσης στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Δύο λόγια τώρα για την καλύτερη υλοποίηση. Η πρόταση ενθαρρύνει την Επιτροπή να είναι ενεργότερη στην χρήση των υφιστάμενων εξουσιών για την επιβολή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αντισταθεί σε οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση και να ξεκινήσει αμέσως διαδικασίες παραβάσεως σε περιπτώσεις όπου μηχανισμοί επίλυσης των ε, προβλημάτων πριν την άσκηση της ένδικης προσφυγής ε, αποτυγχάνουν. Ζητά από την Επιτροπή να μειώσει τις καθυστερήσεις υλοποίησης των οδηγιών τη ενιαίας αγοράς στο 0,5% 20% συμπεριλαμβάνοντας και τις εκκρεμής και τις ανεπαρκείς υλοποίησεις μέχρι το 2012. Επίσης ζητούμε από την Επιτροπή να θέσει ορόσημα 12 μηνών για, την μέγιστο, για το μέγιστο ε, μέσο όρο για την, διαδικασία παραβα... για την διαδικασίας παραβάσεων από τη στιγμή που ε, ανοίγει ο φάκελος τη στιγμή αποστολή της αίτησης στο δικαστήριο. Ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα χρονικό όριο για τη συμμόρφωση των μελών στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά την καλύτερη νομοθεσία, την καλύτερη ρύθμιση τώρα, προτείνουμε η χρήση της, ε, των κανονισμών και όχι των οδηγιών θα συμβάλλει σε καλύτερο, σε σαφέστερο ρυθμιστικό πελαίσιο και θα μειώσει τι δαπάνε συναλλαγή που συνδέονται με την μεταφορά τη νομοθεσία. Επίση, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να παράσχουν πίνακε συστήχηση για όλε τι οδηγίε ενιαία αγορά, καθιστώντα τι δημόσια, ε, καθιστώντα του πίνακε αυτέ δημόσια προσβάσιμοι στου πολίτε. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό και την επίλυση προβλημάτων, προτείνουμε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συντονίζουν και όπου είναι ενδεδειγμένο να ενοποιήσουν τις ε, πολυάριθμες μόνο απευθυντικέ υπηρεσίες για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων. Επίσης ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να καταστήσουν, να δημιουργήσουν σημεία ενιαίας επαφής με βάση την, υπηρεσία, την οδηγία της υπηρεσια πραγματικα πραγματικά one-stop shop με όλες τι πληροφορίε για τι ε, δραστηριότητε των επιχειρήσεων. Κλείνω με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Υπογραμμίζουμε την αμοιβή αξιολόγηση που προβλέπεται στην οδηγία υπηρεσιών ως καινοτόμο τρόμο χρήση ε, τη πίεση από ομολόγου για τη βελτίωση τη ποιότητα τη μεταφορά. Υποστηρίζουμε όπου είναι δεδειγμένο την χρήση τη αμοιβή αξιολόγηση και σε άλλου τομεί. Όπω για παράδειγμα ο τομέα τη ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα εργασία. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 7η Φεβρουαρίου προτιθέμεθα να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες με τους σκιώδεις συζητητές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στην επόμενη σύνοδο στο, ε, στην Ολομέλεια 14 και 17 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο και να γίνει και μια άλλη συνάντηση μεταξύ των τριών εισηγητών πάλι στις 17 Φεβρουαρίου. Αυτά και ευχαριστώ πρόεδρε. Uh, thank Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή Αντώνιο Κόρε Αντεκάμπος για να παρουσιάσει το δικό του κεφάλαιο και ο κύριος Βίζο επίσης, οπότε ελπίζω και αυτός να έρθει εκεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους σκιώδης εισηγητές για αυτή την έκθεση καθώς επίσης και τους ε, Άλλου εισηγητέ ε, για τι συνεδριάσεις και τον συντονισμό που ήδη είχαμε και όπου όπω αναφέρθηκε από την κυρία πιο πριν ήταν όλα αυτά πήγαν πολύ καλά. Πιστεύω ότι θα έχουμε χρόνο για, και πολύ χρόνο, ε, περιθώριο χρονικό για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και να συζητήσουμε καλέ τροπολογίε Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ε, πράξη για την ενιαία αγορά και την κοινωνία, η οικονομία της ε, ε, αγοράς που θα είναι ανταγωνιστική είναι αυτό που αναλύθηκε από κοινού με 19 πρωτοβουλίες όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά. Η έκθεση GREC 2010 είχε προτείνει μια ολιστική σφαιρική αντιμετώπιση για την ανανέωση, ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και την ενεργειακή και βιομηχανική πολιτική και πολιτική για τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση μεταξύ αυτή τη ανακοίνωση και τη ανακοίνωση 2020 ωστόσο δεν είναι απόλυτα σαφή ακόμα. Πρέπει να εργαστούμε για τη συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα και καλύτερη διακυβέρνηση, ώστε η ανανεωμένη, ενδυναμωμένη εσωτερική αγορά να συνεισφέρει για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει εμπιστοσύνη στους ε, καταναλωτέ και πολίτε. Επικεντρωθήκαμε στην αγορά στι μηχανιστικέ εργασίε διεργασίε και πολύ λίγο στι ε, ε, ανησυχίε και τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, των εργαζομένων, πράγμα που μπορεί να επεξηγήσει ένα μέρος ε, του δισταγμού και της κόπωσης των Ευρωπαίων έναντι της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Σημαντικό είναι οι πολίτες να βρεθούν στο επίκεντρο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Τώρα, όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Πρέπει μια εγκάρσια, οριζόντια διάταξη να εισαρθεί η ενιαία εσωτερική αγορά Πρέπει να επιβεβαιώσουμε το άρθρο 9 της Συνθήκης Λισαβόνας και τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι πολιτικέ που θα αναπτυχθούν να επικεντρώνονται στου πολίτες. Να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, να διασφαλίσουμε τη συνοχή μέσω πλήρους ε, σεβασμού των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε το καθήκον από πλευρά Επιτροπή ε, να, ε, να, εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η επίπτωση στην εσωτερική αγορά κάθε πρωτοβουλία. Το γεγονό ότι η Επιτροπή δίνει απαντήσει σε σχέση με το νομοθετικό έργο για την εισαγωγή βεβαιότητα νομική και ασφάλεια για τι υπηρεσίε γενικού ε, συμφέροντο είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με την συνθήκη Λισαβόνα που δίνει μια νέα νομική βάση για αυτό το στόχο. Η πράξη για την ενιαία εσωτερική αγορά πρέπει να έχει στο επίκεντρο τι υπηρεσίε ε, και τα κοινωνικά θέματα και να ληφθούν υπόψη άμεσα τα θέματα με τι δημόσιε συμβάσει και την παροχή υπηρεσιών. Προτεραιότητε προτεραιότητε τώρα. Υπάρχει ανάγκη πρακτικά να καθοριστούν οι προτεραιότητες μεταξύ των 19 αυτών προτάσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η επιλογή να βασίζεται σε πέντε αξίες την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πολιτών, την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπαραγμάτων, ε, τα κοινωνικά θέματα, τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ενίσχυση εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς. Πρακτικά αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν για τους πολίτες. Καθορισμός ε, των προτεραιοτήτων σε κάθε είδους δράση που πρέπει να λαμβάνει υπόψη προτάσεις που θα δίνουν ωφέλη, χειροπιαστά ωφέλη για τους πολίτες και καταναλωτές. Δηλαδή χειροπιαστός συγκεκριμένος, εξειδικευμένος τρόπος παρέμβασης μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο περίοδο και βιωσιμότητα είναι αναγκαίο να υπάρξει έλεγχος και ε, αξιολόγηση για τις επιπτώσεις. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα ε, απόλυτα. Πρέπει να αξιολογήσουμε την ταχύτητα και δυνατότητα, το εφικτό της υλοποίησης αυτών των ε, μέτρων σε σχέση με το 2011. Και μια και δεν έχουμε ακόμα αυτά τα μέτρα, ταυτίζουμε, εντοπίζουμε πέντε τομείς δραστηριότητα το 2011. Πρώτον, ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στις υπηρεσίες, δημιουργώντας μια ενιαία εσωτερική αγορά που θα είναι ε, ολοκληρωμένη για να ξανατεθεί το θέμα της ε, λειτουργικότητας και να αρθούν τα ε, τραπεζικά εμπόδια και προσκόμματα και φορολογικά εμπόδια. Δεύτερον, γοργά να καταλήξουμε σε μια δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να διευθετηθούν τα θέματα και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτόν. Τρίτον, ένα πρόγραμμα δράσης κατά των προϊόντων απομίμησης, προϊόντων μαϊμούδων και προληπτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα όσα θα κυκλοφορούν στην ενιαία εσωτερική αγορά δεν θα αποτελούν κίνδυνο για την κατανάλωση και θα ανταποκρίνονται σε ρήτρε και ε, διατάξει ε, ασφαλή. Τέταρτον, μια πολιτική για την επικοινωνία αποτελεσματική για την πράξη για την ενιαία εσωτερική αγορά, εποπτεύοντα ε, το τι θα συμβαίνει με του πολίτε. Και δείκτε, τέλο, ορόσημα για τα οριζόντια αυτά μέτρα, λαμβάνοντα υπόψη όλα τα μέτρα στην ενιαία εσωτερική αγορά όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις, την εξειδικευσή και δυνατότητα να έχουν αποτέλεσμα δίνοντας απαντήσεις στην ενιαία εσωτερική αγορά και τις ανάγκες για τους πολίτες. Εργάστηκα στενά με τους κοιόδης εισηγητές κυρίες και κύριοι, με ε, τον κύριο Μπουσόη και την κυρία εισηγήτρια. Πιστεύω έτσι ότι μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας σε σχέση με το Συμβούλιο, την Επιτροπή, με τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου για τις δυνατότητες που θα έχουμε για την ενιαία εσωτερική αγορά λαμβάνοντας υπόψη συμμετοχή των πολιτών, λαμβάνοντα υπόψη και τη συμμετοχή, ε, ενεργό συμμετοχή και των επιχειρήσεων. Και έτσι λοιπόν με αυτή την έννοια ε, θα υπάρξει συνένεση ελπίζω και για αυτού του τρει τομεί που θα είναι κοινοί τομεί για όλε τι εκθέσει και θα επιτρέπουν μια ευανάγνωστη δυνατότητα αυτή τη ε, εύληπτη αποδοχή αυτή τη έκθεση με ευανάγνωστο τρόπο. Restoring confidence, αποκαθιστώντα την εμπιστοσύνη, θέτοντα του πολίτε στο επίκεντρο, στην καρδιά τη ενιαία εξωτερική Επίσης θέλω να αναφέρω αυτές τις πέντε προτεραιότητε, που είναι η, η καρδιά αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Ah, Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο εισηγητές. Ο κύριος Μισό ακόμα δεν έχει έρθει, οπότε αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να περάσουμε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής και τους επισκέπτες. Ο κύριος Σίμψον λοιπόν θα μιλήσει για τις ε, πτυχές που επηρεάζουν την έκθεση Μπιζόη και φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα κρατήσουν σημειώσεις και θα του τα διαβιβάσουν. Έχετε λοιπόν το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας πω πως ε, εκ μέρου ε, τη Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Είμαστε ευγνώμονε για τη συντονισμένη προσέγγιση που ακολουθήσατε για τι εκθέσει που ακολουθούν την ανακοίνωση τη Κομισιόν για την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν για την ενιαία αγορά. Όπως ξέρετε, η ανακοίνωση της Κομισιόν σκοπεύει να δώσει όθηση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, κάτι το είναι σημαντικό εάν είναι να ανακάμψει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την οικονομική κρίση και επίσης να δείχνουμε σε μελλοντική ανάπτυξη και ελευθεριστικότητα. Επίσης, μου δίνει τη ευκαιρία να τονίσω την σημασία του τομέα των μεταφορών σε όλα αυτά. Και βεβαίως ε, η ενιαία αγορά ε, και η διακίνηση αγαθών ε, και ανθρώπων εξαρτάται από τις μεταφορές επίσης οι μεταφορές είναι στο μέσο που δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει απασχόληση όχι μόνο μέσω της ε, παροχής υπηρεσιών μεταφορών αλλά και με την κατασκευή οχημάτων και συστημάτων κάθε ε, τρόπο μεταφοράς. Εμείς λέμε στην Επιτροπή μας πως ε, ασχολούμαστε από το ποδήλατο μέχρι το ΤΖΒ και από ένα κάρο που σέρνει άλογο μέχρι το Airbus 380. Όπως λοιπόν ε, λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, οι μεταφορές είναι το νευρικό σύστημα ολόκληρης της οικονομίας. Ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών έχει ουσιαστική σημασία για ανθρώπους, υπηρεσίες και αγαθά. Οι ουσιαστικές ε, ελευθερίες βεβαίως ε, που θεωρούμε σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς. Αλλά ακόμα απέχουμε από μια ενιαία αγορά στον τομέα των μεταφορών και δεν, δεν μπορώ να τονίσω αρκετά το οικονομικό κόστος που έχει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη δει τα ωφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της ε, κοινή αγοράς στον τομέα της αεροπορίας. Υπάρχει λοιπόν η ίδια δυνατότητα για τον τομέα των σιδηροδρόμων και των οδικών μεταφορών και θα επιφέρει αυτό σημαντικές μειώσεις του κόστους. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως τις δυσκολίες δημιουργίας ενίας αγοράς σε κάποιους από αυτούς τους τρόπους μεταφορών, ειδικά στους σιδηροδρόμους, αλλά αυτό δεν ε, μας αποθαρρύνει από τις προσπάθειές μας για να καλύψουμε και αυτόν τον τομέα. Έχουμε ήδη δει τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη μείωση του κόστους ε, μεταφοράς ε, φορτίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ενιαίας αγοράς. Το να δημιουργήσουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των λιμένων και των ε, ποτάμιων μεταφορών επίσης θα έχει έναν αντίκτυπο. Αυτά Βεβαίω θα εξεταστούν στη μελλοντική Λευκή Βίβλο τη Κομισιόν ε, για τις μεταφορές που θα προταθούν μέτρα για να μειωθούν ε, τα εμπόδια μεταξύ διαφόρων μέσων μεταφορά και εθνικών συστημάτων μεταφορών. Επίσης θα υπάρξει και η ανακοίνωση της Κομισιόν για τον νόμο περί ενιαίας αγοράς που κάνει δύο συγκεκριμένες προτάσεις για τον τομέα των μεταφορών που θα ήθελα το Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής σας να αναφέρει στο ψήφισμα. Πρώτη αναφορά είναι η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η Επιτροπή μου θέλει να τονίσει πως οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές θα πρέπει να απομακρυνθούν από μια σειραφή εθνικών έργων αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή, σε πράγματα που έχουν πραγματικά ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, όπως ε, αναγνωρίζει και η στρατηγική για το 2020 που ορίζει την ε, αξία στρατηγικών έργων τα οποία αφαιρούν ε, στενοπούς ειδικά όταν είναι διασυνοριακά και πάντα τονίζουμε τον σημασία του διαδρόμου Περπινιών Περπινιών-Βαρκελών και οι Ισπανοί συνάλφοι θα το γνωρίζουν. Μια ωραιότατη ε, γραμμή σιδηροδρόμου Μαδρίτη-Βερολίνο, το ίδιο επίσης Παρίσι-Περπινιάν, αλλά τίποτα στο ενδιάμεσο. Οπότε πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε εκείνα τα έργα τα οποία έχουν περισσότερη προστάμενη αξία και να διασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Γι' αυτό, στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή μας θέλει να υποστηρίξει την έννοια ενός δικτύου πυρήνα με κάποια βασικά έργα που τηρούν αυτές τις αρχές. Τα έργα αυτά κατόπιν θα πρέπει να είναι η βασική δικαιούχοι στήριξης, επένδυσης και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συνδεθούν με τις τα άλλα έργα σιδηροδρομικών υποδομών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Η δεύτερη αναφορά στον νόμο περί εσωτερικής αγοράς αφορά τα δικαιώματα επιβατών που έχουμε τώρα για όλες βασικές μορφές μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη φάση των δικαιωμάτων επιβατών, θέλουμε η Κομισιόν να δώσει μια γενικότερη κατεύθυνση για τα χρόνια που έρχονται ειδικά, να δει το πώς θα οικοδομήσουμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε και ποιες αδυναμίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η Επιτροπή μου θα ήθελε να σας πει, να τονίσει την σημασία αναθεώρηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων επιβατών, ειδικά όταν μιλάμε για τον τομέα της αεροπορίας, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πού χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις και να είμαστε ειλικρινείς για το πού πρέπει να κλείσουν παραθυράκια. Οπότε πώς θα διευκολύνουμε περισσότερο την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων εντός ενίας αγοράς. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα πρέπει να ακολουθεί από νομοθετικές προτάσεις για να ενισχυθούν και να διευκρινιστούν αυτά τα δικαιώματα, για να υπάρχει ενιαία εφαρμογή, για να μην υπάρχει κίνδυνος στρέβλωση του ανταγωνισμού και εντός των μέσων μεταφοράς και μεταξύ αυτών. Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε τα πακέτα, τα τουριστικά, τις χρεοκοπίες, έχουμε ακούσει χρεοκοπίες αεροπορικών εταιριών και τις υπερβολικές χρεώσεις για υπηρεσίες όπως παραδείγματο χάρη χρέωση για χρήση της τουαλέτας που θα ήθελαν να μας επιβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες. Κύριε Πρόεδρε, καταλήγοντας, θα έλεγα θα σας ε, πρότεινα εξ ονόματος της Επιτροπής μου η δική σας Επιτροπή να συμπεριλάβει τις παραγράφους σας έχω αποστείλει γραπτός στο σχέδιο ψηφίσματος για να μπορέσουμε όπως ε, θεωρούμε να παίξουν οι μεταφορές ε, τον ρόλο τους στην εσωτερική αγορά ένα ρόλο απολύτως κρίσιμο εάν είναι να έχουμε μια στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 ή οποιαδήποτε άλλη στρατηγική να υλοποιηθεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως είπα στην αρχή, για την ευκαιρία που μου δώσατε, μας δώσατε να εμπλακούμε και για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω να εκπροσωπήσω την Επιτροπή μου εδώ πέρα σήμερα. Θεωρώ πως είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα που η Επιτροπή μας είπε πως πρέπει να έρθει ο πρόεδρος της εδώ πέρα, ο υποφαινόμενος δηλαδή, και βεβαίως ως καλός δημοκράτης εκπλήρωσα την εντολή που μου έδωσε η Επιτροπή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, uh, Brown, Πρόεδρος, πρέπει να πω ευχαριστώ πολύ πραγματικά εναντιμών για αυτή την πολύ σαφή τοποθέτηση αμφωτέρων των θεμάτων που αναφέρεται που έχουν τεράστια σημασία και που ουσιαστικά στην έκθεση του κυρίου Κορέντε Κάμπος ε, αναφέρονται. Ε, να τον καλέσω να τοποθετηθεί σύντομα σε αυτά που είπατε. Γνωρίζω ότι με συμπάθεια θα γίνουν αποδεκτά και ως ε, σκιώδης αναφέρομαι, αλλά και ευρύτερα. Σας ευχαριστούμε για το ότι ήρθατε. Αυτό δείχνει την αξία αυτής της πράξης για την ενιαία εσωτερική αγορά συνολικά αναβαθμίζοντας σημαντικά θέματα και καθιστώντας δυνατές πολιτικές όπως για τις μεταφορές και ομιλώ και εξ ονόματος όλης νομίζω της Επιτροπής εδώ λέγοντας ότι δεν έχουμε ενσωματώσει τις ε, πολιτικές μεταφορών επαρκώς ε, στο πλαίσιο και των εγχειρηματών και των φιλοδοξιών για την πολιτική, για την στατική, για την πολιτική 2020 συνολικά. Δεν είχαν πραγματικά αναβαθμιστεί αυτά τα θέματα μεταφορών σε αυτή την πολιτική και τα αιτήματα που συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πράξη για την εσωτερική αγορά ήταν να προσπαθήσουμε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών να διασφαλιστεί, διότι όπως αναφέρατε η εσωτερική αγορά δεν θα επιτύχει πλήρως το δυναμικό της χωρίς τα ε, θέματα μεταφορών που πρέπει να ενταχθούν στα άλλα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια καλή γνωμοδότηση για, για μια άλλη ακόμα λευκή βίβλο για την, ε, τα θέματα μεταφορών ε, που με αφοπλιστική ε, θα έλεγα ε, με αφοπλιστικά τακτό χαρακτήρα εμφανίζονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την προθυμία σας και για το πακέτο για τα τη μετακίνηση και τα ταξίδια. Ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή και για τα θέματα που θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν σε σχέση με τους συντονιστές. Ο κύριος Κορέντε Κάμπος, να απαντήσετε μια και η δική σας έκθεση αφορά και τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από τον κύριο Σίμψον και μετά τον κύριο Μπουσόη θα καλούσα να λάβει τον λόγο να δοθεί συνέχεια σε αυτά. Νομίζω κύριε Κορέντε σαν, σαν, καλό θα ήταν να δίνατε μια απάντηση. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Σίμψον. Είναι χαρά να σας συναντούμε υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και πραγματικά σας ευχαριστούμε γιατί είσαστε παρόν διότι φυσικά θα μπορούσατε να μας αποστείλετε αυτές τις σημειώσεις ε, και με τον κομψό τρόπο, αλλά η παρουσία σας αυτή είναι πολύ πιο ε, εμπλουτιστική και πιο σημαντική για να μπορέσουν αυτές οι προτάσεις ε, να τονιστούν. Να υπογραμμίσω ότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και την χώρα από την οποία προέρχομαι, την Πορτογαλία, για την σημασία των διευρωπαϊκών <clears throat> δικτύων μεταφορών και σε σχέση με τις σημερινές αναφορές. Δεύτερον, για τα δικαιώματα των επιβατών. Θεωρούμε <clears throat> ότι είμαστε μάρτυρες κατά τα τελευταία 5 ε, και 10 ε, χρόνια τεράστιων ε, αλλαγών, επαναστατικών μεταβολών όσον αφορά και τα, τους σιδηροδρόμους. Και φυσικά δεν έχουν όλα ολοκληρωθεί ακόμα και πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα επιβατών με χειροπιαστό πρακτικό τρόπο και λαμβάνοντα υπόψη και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Πρέπει να συγκεραστούν και τα δύο δικαιώματα επιβατών και επιχειρήσεων. Για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων επίσης ένα ουσιώδες στοιχείο το οποίο προσπαθούμε να διασφαλίσουμε και όλο και περισσότερο ανησυχούμε για το θέμα των bailouts και των υπερβολικών κομίστρων και ε, τελών και σε σχέση με κάθε χώρα αυτό το βλέπουμε πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές σας ε, για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε σχέση με όλα αυτά. Και εν τέλει, και προσβλέπω το να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να δούμε τις ε, συστάσεις ε, που θα διαβιβάσετε στο ΜΑΚΟΝ. Δεν ξέρω αν έχουν διαβιβαστεί ήδη αυτές οι προτάσεις σας, οι συστάσεις σας. Δεν έχουν φτάσει ακόμα. Είναι η απάντηση προς τον κύριο Κορέα. Ναι, προσβλέπουμε να δούμε ποιε θα είναι οι συστάσει και θα ληφθούν πλήρω υπόψη. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στη συνέχεια τώρα και θα ακούσουμε από τον τρίτο εισηγητή μα κύριο Μπουσόη, Κριστιαν Μπουσόη και θα αρχίσει και ο γύρος τι παρεμβάσει. Αν θέλετε λοιπόν κυρία Κρατσερμπίρτ να αναφερθείτε σε αυτά Ρούλο Κρότσμαν και οποιοδήποτε άλλο θέλει να προσθεθεί το όνομά του σε αυτόν τον γύρο, Στάιλερ, και η κυρία Γκέπχαρντ και η κυρία Τούνεσε Λεκεγκάρντ Υποθέτω ότι όλοι σας θα θέλετε να εγγραφείτε στον κατάλογο εκείνων που θα παρέμβουν. Λοιπόν, ας ακούσουμε από τον κύριο Μπουσόη πρώτα τα σχετικά που είναι ο τρίτος εισηγητής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ενιαία εταιρική αγορά αναμφισβήτητα είναι ένα μείζον εγχείρημα και ήταν ένα κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όμω η λειτουργία τη ενέργεια εσωτερική αγορά μπορεί να βελτιωθεί. Χρειάζεται διαρκώ προσαρμογέ και εμβάθυνση για να ανταποκρίνονται καλύτερε ανάγκε των καταναλωτών, πολιτών και επιχειρήσεων. Όλοι υποστηρίζουμε τον ρόλο των επιχειρήσεων για την οικονομική ανάκαμψη και την ε, μελλοντική μας οικονομική ανάκαμψη. Γι' αυτό η αναζωογόνηση αυτής της προσπάθειας πρέπει να λάβει υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτό είναι προϋπόθεση για την αποκατάσταση εμπιστοσύνη ε, των πολιτών στην ενιαία εσωτερική αγορά. Μετά, ξεκινώντα την ενιαία εσωτερική αγορά, σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Συνεισφέροντα την ανταγωνιστικότητά του, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διασύνδεση μεταξύ τη πράξη για την την ενιαία εσωτερική αγορά και τη στρατηγική για το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σχέδιο έκθεση καθορίζω τέσσερι τομεί προτεραιοτήτων για να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο. Πρώτον, η ενιαία εσωτερική αγορά πρέπει να, γίνει ένα καλύ... να δημιουργήσει ένα καλύτερο πλαίσιο για καινοτομία. Πρέπει να είναι ο κινητήρα για την ευφυή e και αηφόρο ανάπτυξη. Όλοι ονειρευόμαστε για ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή κοιλάδα Silicon Valley. Αλλά πρέπει να ληφθούν εκείνα τα εγχειρήματα, οι πρωτοβουλίε για να συνεισφέρουμε σε αυτό. Προστασία ιδιωτικό, ε, πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών είναι ε, και αυτό ένα σημείο που έχει ρόλο κλειδί να διαδραματίσει. Επίσης ελπίζω ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν σε αυτό το εγχείρημα. Πρόσβαση στην χρηματοδότηση για την καινοτομία έχει μεγάλη σημασία νέα ε, τέτοιου είδους ε, προγράμματα θα έχουν ε, αποτελεσματικό ρόλο για να διαδραματίσουν σε σχέση και με την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους. Πρέπει να δούμε ότι ο κύριος στόχος είναι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλειών. Πρέπει να δούμε υπό ποιου όρου ε, θα γίνει αυτό όταν θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για αυτόν τον τομέα. Δεύτερο τομέα μια ψηφιακή ενιαία εσωτερική αγορά για τα ψηφιακά θέματα. Έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και συμφωνούμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να προαχθεί για τι διασυνορικές αγορέ. Είναι υποφέλε και για τι επιχειρήσει και για του καταναλωτέ για την ψηφιακή ενιαία εσωτερική αγορά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί και θα έχει περιεχόμενο τα ψηφιακά συνολικά. Να αντιμετωπιστεί το θέμα, το πρόβλημα των προϊόντων απομίμησης και να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνιών. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενός προγράμματος δράσης κατά των προϊόντων απομίμησης. Για τα οπτικοακουστικά και τις υπηρεσίες, αν θέλουμε να προχωρήσουμε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν όλα τα ωφέλη που θα αποκομίσουμε από αυτή τη δράση. Τρίτη προτεραιότητα, τρίτος τομέας θα πρέπει να ληφθούν τα εύθετα σκόπιμα μέτρα για να δημιουργηθεί η ενιαία εσωτερική αγορά με ένα πλαίσιο, με ένα περιβάλλον που θα είναι φιλικό για τι επιχειρήσει. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκε όλων των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίω επειδή λόγω κατακαιρματισμού τη αγορά είναι οι πιο ευάλωτε και λόγω προβλημάτων για την χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα όμω είναι ο κινητήρια, η κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διασφάλιση των θέσεων απασχόληση στο μέλλον. Η βελτίωσή του ε, και η συνδρομή προς αυτέ ε, θα έχει σημαντικό ρόλο. Πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύσσουν το ρόλο τους στην ενιαία εσωτερική αγορά. Μέτρα όσον αφορά την φορολογία που θα ανακουφίζουν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν και αυτά το ρόλο τους. Ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη τον ρόλο των ΜΜΕ διασυνοριακά. Γι' αυτό ένα πιο αποτελεσματικό φιλικό περιβάλλον για αυτές θα πρέπει να, ε, να θεωρήσουμε ότι θα είναι θετικό για τη δράση τους. Θα πρέπει να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια. Τελευταίο το μέσα είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενιαία εσωτερική αγορά για την παροχή υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της ε, ενιαίας εσωτερική αγοράς ε, ιδιαίτερα για τις ε, υπηρεσίες στο διαδίκτυο, μέσω διαδικτύου πρέπει να ενταχθούν στην μέση διάταξη. Αυτές είναι οι υπηρεσίες του μέλλοντος. Εκείνες που θα είναι σύγχρονες και καινοτόμες και χρειαζόμαστε απόλυτα. Και τέλος, σε κατακλείδη θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις τεχνικές πτυχές αυτών των θεμάτων. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που επέλεξα όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα και αν θα ήταν σημαντικό να μπορέσουν και οι 50 προτάσεις να υλοποιηθούν. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μία δέσμη προτεραιοτήτων στην οποία θα επικεντρωθούμε και θα προσθεθεί και ένα νέο πλαίσιο για να λειτουργήσουν αυτές καλά. Τώρα, σε σχέση με την ταυτοποίηση από πλευρά συναδέφων άλλων προτεραιοτήτων, σε σχέση με την ε, ε, ε ανακοίνωση τη Επιτροπή, είμαι πρόθυμο να συζητήσω αυτά τα θέματα με του χειόδη εισηγητέ και τα άλλα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να καταλήξουμε στα βέλτιστα αποτελέσματα. Να έχουμε μια ισχυρή θέση που θα προαγάγει την ενιαία εσωτερική αγορά αποτελεσματικά. Θα ήθελα να πω επίση δύο λόγια για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Συμφωνήσαμε χθε εγώ και οι άλλοι εισηγητέ ότι ε, ποια θα πρέπει να είναι η γενική δομή αυτών των προτάσεων στι εκθέσει. Να προσθεθεί ένα νέο τμήμα ταυτίζοντα, ταυτοποιώντα τα πέντε σημαντικότερα πεδία από όλα όσα αναφέρονται στο σχέδιο έκθεση. Πρέπει να υπάρχει ευρεία συνένεση για το τι θα σημαίνουν αυτέ οι πέντε προτεραιότητε. Συζήτησαμε αυτά σε λεπτομέρειες με τους εισηγητές σε σχέση με την Ολομέλεια του Στρασβούργου το Φεβρουάριο το Φεβρουάριο. Επίσης πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις ε, μεταξύ των ε, προτάσεων στις εκθέσει μας και των θεμάτων. Μια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το εμπόριο στο διαδίκτυο και αυτά τα θέματα αφορούν ε, προτάσεις και οι προτάσεις επίσης του κυρίου Κορέντε Κάμπος για τι τις εμπλεκόμενες αυτές αναφορές καλή ιδέα είναι Επίσης, κάθε ένας από εμά έχοντας ε, συναντήσεις με τους ε, ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να προχωρήσει ώστε να συντονιστεί η δουλειά μας και να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και το σθένος της τελικής μορφής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους τρεις εισηγητές. Τώρα, ας ανακεφαλαιώσουμε για τους ομιλητές και να σας πω ότι προτείνω. Νομίζω πως λογικό είναι πρώτα απ' όλα να αφήσω τους σκιώδεις ηγητές να μιλήσουν, να δώσω το λόγο σε αυτούς και προτείνω να τους ομαδοποιήσουμε με τη σειρά με την οποία ακούσαμε και, τις... και τους ηγητές. Και αν θέλουν να σχολιάσουν μετά από κάθε μπλοκ ομιλητών οι ηγητές βεβαίω έχουν το δικαίωμα. Οπότε θα ακολουθήσουμε την εξής ε, σειρά. Ελπίζω να μην είναι πολύ πολύπλοκα τα πράγματα για την έκθεση Κανιέτη. Λόχιγκαρτ, Ριούλε και Μακλάρκιν είναι όλοι εδώ. Οπότε προτείνω να ακούσουμε πρώτα αυτούς και μετά την κυρία Κανιέτη αν θέλει να σχολιάσει. Μετά για την ε, ενιαία αγορά για τους Ευρώπης έχουμε τον Κρόιτσμαν, εμένα και τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Για επιχειρήσεις και ανάπτυξη Μόνο η κυρία Βανιέο είναι εδώ από τους κοιόδης ηγητές. Εγώ έχω εντολή να εκπροσωπήσω τον κύριο Κουσούσνικ και μετά η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και Χαρτ και Στάιλερ. Αν θέλουν να παρέμβουν μπορούν να μου κάνουν νόημα μετά τους σκιώδης ηγητές. Και θα επανέλθουμε. Νομίζω και η κυρία Ρούλε είπε πως θέλει να μιλήσει και στις άλλες Ωραία. Θα σας προσθέσουμε λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών για να έχουμε έτσι μια δομή για να ακούσουμε και τις τρεις ε, εκθέσεις. Να είμαστε δίκαιοι. Ε, μπορώ να είμαι ευελικτός, αλλά χοντρικά έτσι θα κινηθούμε. Οπότε ξεκινάμε με τα σχόλιά σας και βεβαίω οι σκιώδεις ηγητές μπορούν να αφαιρθούν και σε άλλες ε, εκθέσεις, αλλά κατά βάση στην έκθεση στην οποία είστε σκιώδεις ηγητές. Ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο και Άρτε, επί της έκθεσης κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για να... Ε, first of all, thank you very much, Madam For... πως είμαι σχεδόν ηγητής για την έκθεση περί διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο βεβαίω το υποστηρίζουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πως έχετε συμπεριλάβει τις περισσότερες από τις προτάσεις μου στην έκθεσή σας και θα ήθελα να προσθέσω λίγα πράγματα. Νομίζω πως κάποιες παραγραφή μπορούν να ενισχυθούν και άλλες να προσθεθούν. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να στείλουμε ένα γενικό μήνυμα στην εισαγωγή νομίζω που θα λέει πως χρειαζόμαστε αυστηρή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν ισχύσουμε αυτό το γενικό μήνυμα στην αρχή νομίζω πως θα ήταν καλό. Επίσης μπορούμε να επεκταθούμε λίγο στην παράγραφο 14 ε, το σημείο μια αναφοράς για να ευθυγραμμιστεί αυτή η έκθεση ακόμη περισσότερο με την έκθεση Gephardt για την εφαρμογή της Οδηγίας υπηρεσιών. Θα ήθελα να προσθεθεί μια υποπαράγραφος στην παράγραφο 14 που τονίζει την ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και υπογραφών βασικά αυτά για την παράγραφο 14. Μετά στην παράγραφο 20 για τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών να τονίσουμε το έντονο ενδιαφέρον μας ε, για τους μηχανισμούς αυτούς για τους αλλοδαπούς καταναλωτές θα αυξήσει βεβαίως ε, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα οθήσει το διασυνοριακό εμπόριο. Τέλος να πω πως ε, στην παράγραφο 24 και 25 περί πρόσβαση σε εταίρους κλειδιά και τις εταιρικές σχέσεις. Θέλω να τονίσω πως οι παράγραφοι αυτές έχουν ουσιαστικό ρόλο γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν νομίζω πως η Κομισιόν μέχρι στιγμής ε, ήταν πολύ επιτυχής στην αναδιοργάνωση της εσωτερική αγορά Πρέπει να κάνουμε κάτι. Νομίζω λοιπόν πως παίζουν τον ρόλο κλειδί αυτέ τι παραγραφή και να ενισχύσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Όπως έχουμε συζητήσει τόσες φορές στην Επιτροπή μας, έχουμε πει πω για να ξαναξεκινήσει η οικονομία πρέπει πραγματικά να να το πούμε προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν, την ανάγκη δηλαδή να είναι ακόμη καλύτερη στις προσπάθειές τους. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε έτσι, να έχουμε κάποιες καλές παραγράφους. Αυτά που εμά βεβαίως αναμένω και την συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, πού ήμασταν. Ναι, η κυρία Ρούλε και μετά Μακλάρκιν κύριος Κρότσμαν είπε πως ε, έχει δύο ιδιότητες σήμερα γιατί είναι και εισηγητής για την γνωμοδότηση Επιτροπής Απασχόλησης. Οπότε θα μιλήσει και σε εκείνο το σημείο. Κύριε Ρούλε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το ότι ανέφερε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία συζητήσαμε και έγραψε μια καλή έκθεση η οποία έχει συνοχή και αναφέρει τα σημαντικότερα ζητήματα. Δεν θα αναφερθώ καν σε αυτό το οποίο ε, είπαμε πως θέλουμε να συμπληρωθεί με το Solvit και την ομοθεσία περί ενιαίας αγοράς. Ξέρω πόσο προβληματικά είναι τα πράγματα όταν έχει κανείς πάρα πολύ λίγο χώρο. Δύο πράγματα θέλω να τονίσω ιδιαίτερα και τα δύο αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης της Κομισιόν. Μπορούν να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Το έχω πει πολλές φορές. Αφενός είναι σημαντικό για εμένα η διαδικασία αυτή διαβούλευση να είναι πιο διαφανής γιατί πολλοί από αυτούς συμμετέχουν στη διαβούλευση δεν ξέρουν τι γίνεται με τις απαντήσεις τους, με τις προτάσεις τους και θεωρώ πως η διαβούλευση που θα, για να φτάσει στους πολίτες έχει υποχρέωση να είναι διαφανής και να ξεκαθαρίζει υπό ποια μορφή ε, έχει επεξεργαστεί τυχόν αντιρρήσει Και εδώ πέρα η Κομισιόν μπορεί να γίνει κάπως καλύτερη. Δηλαδή καμιά φορά απορώ με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνουν ε, και έχω σπουδάσει σχετικά και βεβαίως ε, αντιπροσωπευτικό είναι αυτό το οποίο έχει τον υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό καμία φορά το Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η επιστημονική εργασία που γίνεται εδώ πέρα. Και κάτι άλλο θα ήθελα να αναφέρω Κομισιόν στο σημείο 48 στην πρόταση 48 αναφέρει με ποιες ομάδες, με ποιους ενδιαφερόμενους ε, διαβουλεύεται στη διαβούλευση και κάνει διάλογο. Και αυτό το οποίο με κάνει να απορώ είναι το τελευταίο σημείο που μιλάει για τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δεν ξέρω πώς είναι στα αγγλικά, local and regional authorities. Το τελευταίο σημείο στην 48. Α, αυτό δεν είναι. Ε, νομίζω σύμφωνο με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας που έχει ενισχύσει και το ρόλο των Δήμων και της Επιτροπής των ε, Περιφερειών και θα πρέπει νομίζω να αναφέρουμε πως ειδικά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που ασχολούνται περισσότερο με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να συμπεριληφθούν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στην διαδικασία διαλόγου και διαβουλεύσης. Αυτές ήταν οι δύο παρατηρήσεις μου. Ευχαριστούμε κύριε Ρούλε. Κύριε Μακλόκιν. Ευχαριστώ. Και εγώ καλωσορίζω την έκθεση της Κανιέτη για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Πολλές από τις συζητήσεις μας λάβατε υπόψη, παρότι το ότι έχετε περιορισμό στο μέγεθος της έκθεσης. Θέλω να σχολιάσω κάποια σημεία. Οι πίνακε αντιστοίχησης ε, είναι κάτι πολύ θετικό. Δείχνουν ε, βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια. Προσοχή ωστόσο μην χρησιμοποιούμε μόνο κανονισμούς και όχι οδηγίες. Θα πρέπει να υπάρχει και μια κάποια ευελιξία για να καταλαβαίνουμε υπόψη, για να λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές ε, συνθήκες ανακρατών μελών. Ωστόσο υποστηρίζουμε τη χρήση του συστήματος ενίας αγοράς και το One Stop Shop καθώς και την μνήα για τις εναλλακτικές ε, μορφές επίλυσης διαφορών. Εμείς, επίσης, ο μηχανισμός ε, προειδοποίησης που χρησιμοποιούμε στην ε, οδηγία της τις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εδώ. Επίσης, να μειώσουμε το έλλειμμα ενσωμάτωσης που υπάρχει. Χρειάζεται να υπάρξει ισότιμη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη από όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, βασικός παράγοντας αυτό είναι ο εντοπισμός των εμποδίων για να περιοριστούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές. Κατο, τονίζει και η έκθεση. Βεβαίως ο στόχος είναι η σωστά λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Κάθε έκθεση λοιπόν θα πρέπει να ελέγχει κάθε φράση και κάθε τοπολογία για να τηρεί τον στόχο αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήρθε ο κύριος Ραπκάη που είναι υπεύθυνο για την, από σοσιαλιστές αλλά ε, θα σας δώσω μετά το λόγο. Πάντως πρώτα έχει το λόγο ο κύριος Κρόιτσμαν για την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Κανιέτη για το σχέδιο έκθεσης που αποτελεί σημαντική βάση εργασίας. Βεβαίως η διακυβέρνηση στα γερμανικά έχει μεταφραστεί οικονομική διακυβέρνηση και θυμίζει έτσι λίγο κομμουνιστική ορολογία. Ε, δεν νομίζω να είναι αυτό το οποίο ήθελε η εισηγήτρια και οπωσδήποτε αυτό το οποίο θέλουμε φιλελεύθεροι. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ενιαία εφαρμογή των οδηγιών για να έχουμε ασφάλεια δικαίου και μείωση του σχετικού κόστους. Επίσης θα πρέπει να καταρτήσουν πίνακες αντιστοιχεία στα κράτη-μέλη με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής. Επίσης χαιρετίζω τα συγκεκριμένα μέτρα κλειδιά τα οποία αναφέρονται στο τέλος της έκθεσης όπως παραδείγματος χάρη η απέτηση στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή οι πρόεδροι Κομισιών και Συμβουλίου να φροντίσουν για αναζωογόνηση της αγοράς. Μέχρι στιγμής δυστυχώς οι κύριοι Μπαρόσο και Φανρόμπα δεν έχουν πει τίποτα σχετικό. Επίσης καλή ιδέα είναι να δούμε ποια είναι η τωρινή κατάσταση της εφαρμογής των διαφόρων βημάτων των στόχων της εσωτερικής αγοράς και να γίνεται ένας απολογισμός στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Επίσης ε, τονίζω εξ ονόματος Επιτροπής ε, Απασχόλησης ε, πως η ενίσχυση εσωτερικής αγοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες ιδιαίτερα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δουν συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Λοιπόν, η ορθή διακυβέρνηση είναι σωστή, είναι κρίσιμη για να επιτύχουμε την ε, σωστή λειτουργία της εσωτερική αγοράς. Επίσης, όσον αφορά την Επιτροπή Απασχόληση, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η κινητικότητα των εργαζομένων, υψηλό επίπεδο απασχόλησης, ανάλογη βεβαίως προστασία κοινωνική, καταπολέμηση του αποκλεισμού και η βιωσιμότητα των συντάξεων. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέτρα στήριξης έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πολίτες και επιχειρήσεις απαραίτητες πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλα κράτη-μέλη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις δημόσιες αρχές και τονίζω πως χθες είχαμε μια συζήτηση και το ήταν και η κυρία Γκέπχαρτ Και βλέπετε πως ε, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα ενιαία γκισέ ή μάλλον δεν συμβαίνει, δηλαδή αυτό το τίποτα που δεν συμβαίνει είναι ένα αρκετά μεγάλο εμπόδιο και θα πρέπει να έχουμε σημαντική βελτίωση για να γνωστοποιηθούν και αυτοί οι ενιαίοι συνομιλητές, αυτά τα ενιαία γκισέ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει νωρίτερη εμπλοκή των ε, φορέων της ε, κοινωνίας για να γίνουν αντιληπτές πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, να υπάρχει αποδοχή από το λαό και να μην έχουμε πλέον άλλη απώλεια της εμπιστοσύνης. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να ε, προχωρήσει σε ανοιχτό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και όχι να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες. Τέλος, θα πρέπει να ζητήσουμε ιδιαίτερα συμμετοχή από τους κοινωνικούς εταίρους να μιλάμε για νομικές ε, διατάξεις. Γιατί μόνο με κοινέ προσπάθειες θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε αυτό το τομέα. Για το χρονοδιάγραμμα προβλέπουμε 14 Φεβρουαρίου στο... την ψηφοφορία. Ελπίζω λοιπόν να σας ε, βοηθήσουμε έτσι για να περάσει η έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πραγματικά την Επιτροπή Απασχόλησης. Πραγματικά δείχνετε ότι θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας. Από τους Κιώβης, ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, συγγνώμη που ήρθα καθυστερημένα άλλαξε το πρόγραμμά μου τελευταία στιγμή. Γενικά και παρότι δεν μπόρεσα να ακούσω τις πρωινές συζητήσεις, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου με την έκθεση της κ. Κανιέτε. Καλά δομημένη είναι και λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ε, διαστάσεις ε, βελτίωσης της λειτουργίας της ενέργειας αγοράς. Οι προτάσεις της Επιτροπής ήταν επίσης καλές. Τώρα που έχω την ευκαιρία ωστόσο θέλω να ασχοληθώ με κάποια σημαντικά κατά απόψή μου θέματα. Πρώτον, είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστική σημασία και οι πίνακες αντιστοίχησης είναι πολύ σημαντικοί. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί η χρήση τους υποστηρίζω την χρήση αυτών των πινάκων. Κάτι άλλο σημαντικό, το χρονοδιάγραμμα, ώστε τα κράτη-μέλη να απαιτείται να δεσμεύονται ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα ενσωματώσουν και πώς θα ενσωματώσουν τις οδηγίες της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε ε, συγκεκριμένα εργαλεία λειτουργίας. Οι διαδικασίες παραπομπής για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτή θα πρέπει να είναι η βασική μέθοδος αν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πέραν της βελτίωσης της υλοποίησης πρέπει να δώσουμε προσοχή και στην διαφάνεια, στη σαφήνεια και την ποιότητα της, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό είναι πάντα σημαντικό. Οι ασαφείς οδηγίες επιβραδύνουν την ε, εθνική ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και αυτό το καταλαβαίνει και ο πολίτης. Γι' αυτό υπογραμμίζουμε εκ νέου την ανάγκη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών είναι εξίσου σημαντικό με την ανοιχτή νομοθετική διαδικασία για να παράσχουμε ενημέρωση για τα πραγματικά γεγονότα για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε σαφέστερες προτάσεις από την Επιτροπή για το πώς θεωρούν ότι θα διασφαλίζουν το, τη διεύρυνση του διαλόγου με τους πολίτες. Από ό,τι έχω καταλάβει από την Επιτροπή θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες αυτή αντιστοίχησης και άλλες δομές για το στόχο αυτό. Εν γέννη υποστηρίζω τις προτάσεις. Η συνεργασία μεταξύ αρχών και αυτές πρέπει να ενισχυθούν. Η περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος ε, της ε, εσωτερικής αγοράς ε, είναι, των πρωτοβουλειών εσωτερικής αγοράς είναι σημαντικές. Το αναφέρει και η έκθεση Μπουζόη. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η τεχνική εφαρμογή, η μείωση και κατάργηση των νομοθετικών εμποδίων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, βέβαια, πάντα, ότι εδώ είμαστε για να εξυπηρετούμε τους πολίτες και τους καταναλωτές. Δεν θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, διαχείριση και να πολλαπλασιάζουμε τις εκθέσεις. Θα πρέπει να γίνεται αυτό σε ε, επίπεδο βάσης, να λειτουργεί η νομοθεσία σε επίπεδο βάσης η διαχείριση για τα μικρά και τα καινούργια κράτη-μέλη είναι πάντα δύσκολη. Θα πρέπει να, βάλουμε στην, να δώσουμε προτεραιότητα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο χρήσιμε Χρήσιμες παρατηρήσεις. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Η κυρία Κοράτσα Να συγχαρώ την Σάντρα, διότι συμπεριέλαβε όλα τα σημεία που τονίζουμε εμείς στην Επιτροπή την ανάγκη να βάλουμε την πραγματική οικονομία στο κέντρο της μείωσης διάταξης της πολιτικής προσέγγισης, μια ολιστική στάση, μείωση της ε, καθυστέρησης ε, στην ενσωμάτωση και ταχύτερες παραπομπές. Η Επιτροπή είναι η βασική αρμόδια αντιμετώπιση ενίας αγοράς και θα έπρεπε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αναλάβει την πολιτική κυριότητα της επανεκκίνησης της ενίας αγοράς. Μου λείπει ωστόσο εδώ από ό,τι βλέπω ένα αίτημα απορρίθμισης. Θα πρέπει να μιλούμε πάντα για την νομοθεσία για τις μικρές επιχειρήσεις. Η μείωση της γραφειοκρατίας των επιχειρήσεων είναι ένας από τους καλύτερους ρόλους ε, παρότρινσης και ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς και οι συνάδελφοι θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Αγκέπαρντ. Εσείς θέλατε νομίζω να πείτε κάτι σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ακριβώς αυτό το τελευταίο σημείο θα είναι ένα επίμαχο σημείο σίγουρα σε σχέση με τη δική μου ομάδα διότι η απορρίθμιση αυτή δεν μπορεί να είναι απάντηση, αλλά μια λογική σωστή απορρίθμιση, η ίδια η βάση που θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η απάντηση που χρειαζόμαστε σε σχέση με αυτό. Αυτό και πάλι για την τελευταία σας παρατήρηση για αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, πιστεύω ότι για την απορρίθμιση αφεαυτού δεν θα ήταν ε, καλό να βρεθεί στην έκθεση. Εκείνο το οποίο είναι, πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση, ολιστική προσέγγιση όπως ανέφερε ο κύριος Κορέα και για την έκθεση της κυρίας Καλέτε όπου πρόκειται για την καλύτερη διακυβέρνηση και από πλευράς Κρόιτσμαν έχει δίκιο. Τον κομμουνισμό δεν θέλουμε να τον εισαγάγουμε πάλι σε σχέση με την ε, Οικονομική Νομισματική Αυτό θα ήταν η εσφαλμένη προσέγγιση και μετάφραση. Δεν ξέρω με, ποια μετάφραση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, όμως η κομμουνιστική προσέγγιση ήταν, είναι σίγουρα λάθος. Να το δούμε αυτό, κυρία Καλιέτα, είπατε για το σύστημα της αμοιβαία αξιολόγησης, ότι λέει είναι πολύ καλό σύστημα παντού θα πρέπει να εισαχθεί όπου είναι δυνατόν. Εδώ θέτω μεγάλο ερωτηματικό όμως εγώ. Έχω μεγάλα ερωτήματα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα καλό μέσο, ένα καλό εργαλείο. Διερωτώ με όμως, παντού πρέπει να εισαχθεί. Δεν νομίζω. Και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν για την οδηγία περί υπηρεσιών είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ομόφωνα και μετά από πρόταση της δικής σας ομάδας ότι αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση από την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες θέλαμε να την διαγράψουμε. Τα κράτη-μέλη τότε ήθελαν οπωσδήποτε να έχουν μια τέτοια αμοιβαία αξιολόγηση. Και τα κράτη-μέλη είναι σήμερα εκείνα που παραπονούνται και λένε ότι έχει τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση αυτή η ε, προσέγγιση. Σε κάποιους τομείς αυτό μπορεί να είναι θετικό στην περιπαροχή οδηγίας Οπωσδήποτε εκφράζω την ε, άποψή μου σε σχέση με τα όσα είχα, είχα πει πριν από ε, μερικά χρόνια. Πρέπει όμως ε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το μέσο δεν μπορούμε τους υπαλλήλους, ε, τους ε, κρατικούς, ε, τους, τους υπαλλήλους του δημοσίου να τους εξουδετερώσουμε μια και θα τους υποχρεώναμε να συντάσσουν διαρκώς εκθέσεις που θα έπρεπε διαρκώς να αξιολογούνται από τα άλλα κράτη-μέλη και τους υπαλλήλους τους. Δεν μπορούμε έτσι να τους, ας το πω έτσι, παροπλίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να θέσουμε μεγαλύτερη επιβάρυνση, μεγαλύτερη επικέντρωση στις, στους πίνακες αντιστοίχησης ή αναλογίας Γι' αυτό σας παρακαλώ σε σχέση με την έκθεσή σας να το σχετικοποιήσετε αυτό σε σχέση με αυτή την προσέγγιση. Μια και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή είπαμε ότι μια μελέτη θα θέλαμε να συνταχθεί για να αξιολογήσει ακριβώς αυτή η μελέτη τι θα δώσει ως όφελος αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση. Τι θα γίνεται με, τις, με τους πίνακες αντιστήχησης ε, και αναφορό, αναφοράς και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό δεν θα ήταν καλό αυτή τη φάση αυτό το αίτημα με αυτόν τον τρόπο να το διατυπώσουμε όπως το ευρίσκουμε σήμερα στην έκθεσή σας. Είναι μια παρέκκληση που έχω εγώ προς εμάς και θα ήθελα να την λάβετε υπόψη. Ένα δεύτερο σημείο και έχει και αυτό τη μεγάλη σπουδαιότητά του και έχει δίκιο ο κύριος Κρόισμα σε σχέση με αυτό είναι αυτό που εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά και με την οδηγία περιπαροχής υπηρεσιών κάνουμε. Δηλαδή να δούμε επακριβώς και έχουμε και σε σχέση με τα κράτη-μέλη πώς εφαρμόζεται αυτή η οδηγία και όταν πρόκειται για ε, ενιαίους ε, ε, εταίρους βλέπουμε μια, μια καταστροφική κατάσταση. 22 κράτη εισήγαγαν αυτή την υποχρέωση. Σε 17 κάπως λειτουργούν τα πράγματα αλλά για 9 μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα και αυτό δεν είναι καλό. Και τώρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την νομοθεσία αλλά την υλοποίηση, την εφαρμογή και θα έλεγα ότι και εδώ πρέπει εντονότερα να θέσουμε το επίκεντρο στην έκθεση της κυρίας Κανιέτε όσον αφορά την υλοποίηση από τα κράτη-μέλη και την ευθύνη υπευθυνότητα των κρατών μελών όσον αφορά την διακυβέρνηση. Αυτή η διακυβέρνηση ως ε, ευθύνη να εκφράζεται πιο χειροπιαστά, ώστε να βλέπουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για, εθνική, για ευρωπαϊκή πολιτική, ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και για εθνικές πολιτικές που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Και η ε, αντιστοιχία εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών έχει και αυτή τη μεγάλη της ε, σπουδαιότητα. Ευχαριστώ. Για την έκθεση Κανιέτη θέλετε να μιλήσετε. Παρακαλώ. Κύριε Στάιλερ, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Κανιέτη που είναι τόσο συνδεδεμένα όλα τα θέματα μεταξύ τους που είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μία έκθεση μόνο. Το γεγονός ότι για τη νομοθεσία είναι υπεύθυνη εννέα επίτροποι και ότι θα ξεκινήσει η υλοποίησή της ε, στην 20η επέτειο της έναρξης της ενιαίας αγοράς σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση στο τέλος του άλλου έτους. Είναι ρεαλιστικό. Υπάρχουν αυτές οι πέντε προτεραιότητες που είναι πολύ σημαντικές, οι οποίες αφορούν την, ε, το συσχετισμό με τους πολίτες, ε, την διακυβέρνηση για να μπορούν οι πολίτες να καταλάβουν ότι τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και να εξασφαλίσουμε ότι δεν δίνουμε πολλές υποσχέσεις που μετά δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Αυτά που λέμε πρέπει να τα κάνουμε. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Τα προηγούμενα τμήματα της προηγούμενης ε, της ενιαίας αγοράς που υλοποιήθηκαν σωστά ε, είναι, πρέπει να μας βιβάξουν. Η καλύτερη νομοθεσία είναι κάτι που είναι βασικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς, ούτω ώστε να περάσουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι η ενιαία αγορά δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί δουλειές. Αυτό θέλουμε να περάσουμε. Να ρωτήσω λοιπόν την εισηγήτρια, ποια είναι τα πέντε μεγάλα νομοθε... οι πέντε μεγάλες νομοθετικές προτεραιότητες, κατά την άποψή σα. Μίλησε ο κύριος Σίμψον για ορισμένε από αυτές. Αλλά, για παράδειγμα, η ψηφιακή υποδομή είναι κάτι που κατά την άποψή μου πρέπει να υλοποιηθεί. Περιλαμβάνει την ψηφιακή υποδομή στις πέντε μεγάλες ε, προτεραιότητες. Είναι μία από τις μεγάλες προτεραιότητες. Επίσης, λέμε πόσο σημαντική είναι, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Κομισιόν. Ε, όλα τα κράτη-μέλη έχουν περικοπές δημοσιονομικού χαρακτήρα. Μήπως οι προεδρίες θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να βάλουν την ενιαία αγορά στην ατζέντα τους. Το κάνουν, αλλά πιστεύω ότι ως Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο, στους εκπροσώπους Συμβουλίου, λέγοντας ότι το δικό μας όραμα για την ενιαία αγορά είναι να προωθούν αυτή το κείμενο της επιτροπή. Ευχαριστώ. Δύο σχολεία προσωπικά έχω, αλλά δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει να σχολιάσει πριν ε, ολοκληρώσουμε και μετά η κυρία Κανιέτη. Να πω δύο παρατηρήσεις προσωπικά έχουμε στη συνέχεια των παρατηρήσεων του κ. Ρέπος. Αναφέρθηκε στο σύστημα ενημέρωσης της ενιαίας αγοράς. Είχαμε, είχα πάει σε μια διασύνοδο της Επιτροπής, σε μια συνάντηση, μια διάσκεψη που είχε οργανώσει η Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, όπου ήταν πολλοί εκπρόσωποι πολλών δομών και έχω την εντύπωση ότι οι συναντήσεις αυτές δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς από την Επιτροπή. Και κάποιοι άλλοι το είπαν, κύριε Ρούλε. Η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς ε, πηγαίνει συχνά πλέον η υλοποίησή τους δεν είναι εθνική αλλά είναι περιφερειακή τοπική. Μας το είχαν πει αυτό και όταν είχαμε κάνει μια επίσκεψη στη Σουηδία. Η κυρία το αναφέρει στην έκθεση της, ίσως θα έπρεπε να το υπογραμμίσουμε ωστόσο. Και ιδιαίτερα για την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, Φερρυπίν. Οι τοπικές άδειε, οι τοπικέ εγκρίσει αποτελούν μία από τις δυσκολίες που προκύπτουν στην αμοιβαία αξιολόγηση τη οδηγία των υπηρεσιών. Κάποιες ε, χώρες θέλουν να κρατήσουν δικές τους ε, ρυθμίσεις και δικά του ε, δικές τους άδειες για κάποια επαγγέλματα, για την κυπουρική για παράδειγμα, όπου στην ουσία, που στην ουσία συνιστούν μη δασμολογικό εμπόδια. Διάβασα και την έκθεση της Επιτροπής, ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ήθελα να πάω και σε αυτή τη συνάντηση χθες, αλλά δεν πήγα γιατί το, το αεροπλάνο μου από τον Μπέρμιχαμ καθυστέρησε 6,5 ώρες και δεν μπόρεσα να πάω. Ήταν η κυρία Γκέπχαρντ εκεί και διαφύλαξε την ε, παρουσία της Επιτροπής σε αυτή τη συνάντηση. Η αμοιβαία αξιολόγηση ωστόσο είναι σημαντικό. Η κυρία σωστά είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η αμοιβαία αξιολόγηση όπως ενδείκνυται. Σωστή ορολογία. Αλλά κάτι που θα πρέπει να κοιτάξουμε περαιτέρω είναι να γίνει πολύ πιο διάφανη διαδικασία. Δεν είναι σαφές σε μας και στους πολίτες νομίζω ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στις αξιολογήσεις. Γιατί τα κριτήρια αυτά δεν είναι δημόσια, δεν είναι σαφή. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τη διαδικασία αλλά με μεγαλύτερη διαφάνεια στο μέλλον. Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται ορισμένα κριτήρια θα πρέπει να συζητηθεί ε, στο δημόσιο βήμα. Και εμείς είμαστε ένα τέτοιο δημόσιο βήμα σαν Επιτροπή. Δεν ξέρω κάποιο άλλο θέλει να σχολιάσει. Αλλιώ να ζητήσω τον κύριο Μπράμπτεντ να πει δύο πράγματα και να μας διαφωτίσει για την άποψη της Επιτροπής για το ζήτημα που ανέφεραν πολλοί ε, Γερμανοί συνάδελφοι την μετάφραση δηλαδή του όρου στα γερμανικά. Σίγουρα θα έχετε και κάποιο, κάποια σχόλια να κάνετε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε δύσκολο αυτό το εγχείρημα το οποίο μου επομίζεται να βρω τη σωστή ε, μετάφραση για αυτό τον όρο. Δυστυχώς δεν έχω την ε, έκδοση στα γερμανικά του SMA, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθουμε και να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να δώσουμε στη γραμματεία τη σωστή, το σωστό όρο για την διακυβέρνηση Επίσης ε, ευχαριστούμε και την κυρία Κανιέτα για την έκθεσή της ε, και για το πώς τονίζονται τα θέματα αυτά στην προσέγγιση της. Γενικά βλέπουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό ότι προσοχή και προσπάθεια δίνεται στην ε, ταυτοποίηση προτεραιοτήτων σε σχέση με τους άξονες που προτείνονται διότι αυτή είναι η πρόκληση ακριβώς για όλους μας που πρέπει να αντιμετωπιστεί, να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα εργασίας μας και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη και την ευρύτερη συζήτηση εστιαζόμενη στα ορθά θέματα. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση και κατά τα τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου θα αναφέρουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα, α, τις απαντήσεις και την ανταπόκριση που ε, έχουμε. Η συζήτηση λοιπόν ε, διευρύνεται στα γαλλικά θα λέγαμε ότι ενδυναμώνεται και διευρύνεται η ένταση της συζήτησης εμπλέκονται και οι τοπικές περιφερειακές αρχές για τη διεξαγωγή στρογγυλών τραπεζών σε περιφερειακό επίπεδο και η Επιτροπή Περιφερειών επίσης και γι' αυτό αναμένουμε προσδοκούμε ότι πολλές προτάσεις θα υποβληθούν και θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου όπου θα αναμένουμε. Είμαστε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε για να φτάσουμε μέχρι τις περιφερειακές και τοπικές αρχές θα στεφθεί με επιτυχία με τις πολλές απαντήσεις και την εμπλοκή πολλών που θα έχουμε και για το ερωτηματολόγιο ε, που έχει ξεκινήσει και έχει ε, διαδοθεί στο διαδίκτυο μέχρι σήμερα περισσότερο πολίτες έχουν απαντήσει 150 τέτοιες ε, απαντήσεις ε, που είχαμε ε, είχαμε από τις, από τις αρμόδιες αρχές η συντριπτική πλειοψηφία είναι όμως από τους πολίτες για τα θέματα τα οποία εθίγησαν τον ρόλο της αμοιβέ αξιολόγησης η κυρία Γκέπαρτ τοποθετήθηκε σε σχέση με αυτό για την χρήση αυτού του μέσου της αμοιβαία αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, πράξη στο νόμο για την ενιαία εσωτερική αγορά ανέφερε ότι θα πρέπει για κύρια πεδία νομοθεσίας ε, να δρομολογηθεί αυτό. Δεν είναι ε, η προσέγγιση μας η χρήση ως γενικού μέσου αυτής της προσέγγισης. Και εδώ σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, για να είμαστε πιο σαφείς σε σχέση με τα κριτήρια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος όταν έχουμε τομεακή εμπλοκή σε τομείς όπου, για παράδειγμα, όταν έχουμε την ε, ε, εκπόνηση πρόσθετων προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, το gold plating, να δούμε πώς θα γίνεται αυτή η επιχρήσωση, ε, η εκπόνηση αυτών των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο. Δεν ισχύει συλλήβδιν λοιπόν αυτό και θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κάθε φορά συγκυρία. Εδώ έχουμε το θέμα αυτό για τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι πρέπει να γίνει. Χαιρετίζουμε την ε, υποστήριξη που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένοντας και μένοντας τα κράτη-μέλη να υποβάλουν πίνακες αντιστοίχησης και να δημοσιεύονται, να δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Τονίζουμε επίση τη διασύνδεση τη ε, νομοθεσία για την ενιαία εσωτερική αγορά και τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 σε υψηλό επίπεδο όπως τονίζει και η κυρία Κανιέτε στην έκθεσή της. Το χαιρετίζουμε αυτό και το βλέπουμε άρρηκτα ως μέσο, μέτρο α, του να υποβάλλονται σε τακτά διαστήματα εκθέσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής 2020 και που τώρα σε τακτά διαστήματα θα γίνεται και που κατά την αιαρινή Σύνοδο του Συμβουλίου θα είναι η ορθή, η σωστή συγκυρία να συζητηθούν τα θέματα για την πρόοδο για την ενιαία εσωτερική αγορά. Και τέλος, σε σχέση με τα όσα γίνονται από πλευράς της Προεδρίας, θέλουμε να διασφαλίσουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα υπάρχει και έντονη σε βάθος εμπλοκή και της ε, νυν Προεδρίας, της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου αλλά και της μελλοντικής της Πολωνικής Προεδρίας. Είναι στόχος να συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά με τις Προεδρίες μέχρι το τέλος του 2020 ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα θέματα θα βρίσκονται πάνω-πάνω στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων τους. Ευχαριστώ. Ούγγρος υπουργό που μας επισκεφτεί την περασμένη εβδομάδα αυτό ακριβώς είπε. Υπήρξε σαφής βέσμευση της Προεδρίας, κάτι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Κυρία Κανιέτη, θέλετε να κλείσετε. Κοιτάξτε, ziņojumam esiet devuši. Δεν υπάρχει ακόμη διερμηνία. Ένα λεπτό παρακαλώ. So, Mr. Chairman. Πρόεδρε, θα έλεγα ότι έχουν μπερδευτεί κάπως. Λυπούμε πρόεδρε, δημιουργήθηκε κάποια μικρή σύγχυση. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα σε αυτή τη συζήτηση και είχα το δικαίωμα να το κάνω. Δεν, νομίζω ότι οι διοικητικές δυσκολίες δεν νομίζω ότι οι διοικητικές δυσχέρειες είναι μια δικαιολογία, ένα πρόσχημα που θα παρακολουθήσουν τη συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που είμαι πλήρες μέλος εγώ, να μπορώ να παρέμβω στην ε, μητρική μου γλώσσα. Και το γεγονός ότι, πώς να το πω, ότι έχω κάποια ικανότητα να εκφράζομαι σε άλλες γλώσσες δεν δικαιολογεί την ε, απουσία της δυνατότητας να εκφράζομαι στη μητρική μου γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι την επόμενη φορά δεν θα αντιμετωπίζω μια παρόμοια κατάσταση και θα μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα μου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλα τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση παρεμβαίνοντας ε, επί της έκθεσής μου. Ιδιαίτερα αξιολογώ και εκτιμώ όλες τις προτάσεις που κάνατε για τη βελτίωση της έκθεσής μου. Και ο κύριος όρος που μου αρέσει ως λέξη πρακτικά σε όλες τις προτάσεις σας ουσιαστικά είναι η ενίσχυση, η ενδυνάμωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς με κάθε τρόπο, με την υλοποίηση με την καταπολέμηση ε, των παρεκκλήσεων και παραβιάσεων, τονίζοντας τις δράσεις και από πλευράς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα λοιπά και τα ούτω καθεξής. Θα προσπαθήσω τώρα στη συνέχεια να απαριθμίσω και να τα πάρω με τη σειρά όλα τα όσα είπατε εξειδικευμένα. Συμφωνώ με τον κύριο Λόκεγκαντ όσον αφορά την υποπαράγραφο για το σημείο 14 γιατί και εγώ η ίδια στις δικές μου τροπολογίες στοχεύω να τονίσω τον ρόλο του κοινωνικού δικτύου για παράδειγμα του διαδικτύου και με βάση αυτά τα μέσα και δυνατότητες συμμετοχής για τις ανταλλαγές απόψεων και προαγωγή της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό ε, επίσης εφαρμόζεται και για το διαδίκτυο, για την πύλη, την ε, ιστοπύλη για την ενιαία εσωτερική αγορά. Από την άλλη πλευρά, να αναγνωρίσουμε και το ρόλο του, της πύλης Solvit και για τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Και τρίτη ε, προσέγγιση σε σχέση με τροπολογία για τους συναδέφους και πρέπει να αξιολογήσουμε προτάσεις για την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων, εναλλακτικών δυνατοτήτων και της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στο φόρουμ ως δυνατοτήτων που σε τακτά διαστήματα θα αξιολογούν τις εξελίξεις, εξελίξεις στην ενιαία εσωτερική αγορά. Τώρα στη συνέχεια και εν μέρει απήντησα ήδη στην κυρία Ρούλε. Επίσης θεωρώ ότι η διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους ε, Ευρωπαίους ε, και Επίσης, ο ρόλος των τοπικών αρχών για την προαγωγή της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πρέπει να ενδυναμωθεί στην έκθεση. Όσον αφορά την κυρία Μακλάκιν, Πράγματι, με ικανοποιεί το γεγονός ότι υποστηρίζεται την ανάγκη να υπάρχει ε, η ανάγκη της αντιστήχησης των πινάκων αυτών και αυτό πρέπει πραγματικά να ληφθεί υπόψη. Ήδη στην Λετωνία το ε, είδαμε. Η Λετωνία είναι κατά της ε, χρήσης αυτών των πινάκων αντιστάθμισης και αντιστήχησης, με συγχωρείτε. Αληθεύει ότι σε σχέση με τις περισσότερες διατάξεις ε, και ε, οδηγίες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα ρυθμίζουμε αυτά τα θέματα. Είναι όμως σημαντικό να συμπεριλαμβάνετε, να προβλέπετε μια τέτοια προσέγγιση στην έκθεσή μας για αυτούς τους πίνακες αντιστοίχησης. Ευχαριστώ την κυρία Μακλάκιν επίσης για το γεγονός ότι επιβεβαίωσε την εντύπωση που είχα αποκομίσει ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε με άλλα λόγια τον ρόλο των κρατών μελών στην ε, υποχρέωση που υπάρχει να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται οι διατάξεις αυτές μέσα σε σαφή χρονοδιαγράμματα, σαφή χρονοπλαίσια. Γι' αυτό αναφέρω στην έκθεσή μου τις βέλτιστες προδιαγραφές, benchmarking που πρέπει να ισχύει. Τώρα, στη συνέχεια, η τελευταία μου παρατήρηση επιβεβαιώνει αυτό που είπατε εσείς συνάδελφε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην εφαρμογή και υλοποίηση από τα κράτη-μέλη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ε ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κρότσμαν που αφορά, αναφέρθηκε στο τμήμα της έκθεσής μου σχετικά. Χρειαζόμαστε όμως εξίσου αλλά δεν είναι αυτός ο όρος. Ευχαριστώ για το ότι υποστηρίζετε περισσότερο κανονισμούς και όχι τόσο οδηγίες. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μένα προσωπικά. Αλλά είναι τέλος έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να επιλεγεί η σωστή διατύπωση ώστε να παραμείνει αυτό στο σωστό πλαίσιο στην έκθεση θα ήθελα να υπάρξουν περισσότερες συζητήσεις ε, με την κυρία Κοράτσα Μπίλντ όσον αφορά την απορρίθμιση και το τι θα κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τα συναφή θέματα. Ευχαριστώ την κυρία Γκέπχατ και την ευχαριστώ σε σχέση με τις σκόπιμες παρατηρήσεις ε, για την αξιολόγηση, αμοιβαία αξιολόγηση που ε, απορρέει και από την προσωπική της εμπλοκή και συνεισφορά σε αυτό το θέμα και την υποστήριξη των πινάκων αντιστοίχησης. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα καλό θετικό αποτέλεσμα μέσω της έκθεσής μας. Πράγματι είναι σημαντικό πώς υλοποιούν ε, τα κράτη-μέλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα δύο θέματα που έθιξε η κυρία Στάιλερ Ποιε είναι για τις πέντε αυτές προτεραιότητες. Εγώ προτείνω σχετικά προσωρινά, προτείνω επτά τέτοιε προτεραιότητε. Γνωρίζω όμω ότι συνολικά πρέπει να καταλήξουμε στο τέλο τέλο σε πέντε συν πέντε συν πέντε από πλευρά μα. Γι' αυτό είναι δική μα δουλειά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Είμαι πρόθυμη να ακούσω τις προτάσεις σας με ανοιχτό πνεύμα όπως είπα, εγώ θεωρώ την ψηφιακή ημερήσια διάταξη, το ψηφιακό θεματολόγιο ως ε, θέμα προτεραιότητας. Και με αυτή τη βάση θα πρέπει να προσεγγιστεί το θέμα τροπολογιών. Μάκομ Χάρμπορ, έχετε δίκιο σε σχέση με την έλλειψη συγκεκριμένου, ε, συγκεκριμένων στοιχείων επί ε, πτυχών της ενιαίας αγοράς συνολικά. Διότι δημιούργησε σύγχυση, δηλαδή πράγματι εξεπλάγει όταν είδα πόσα stop shops υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό προτείνω να αξιολογήσουμε πρώτα την κατάσταση όσα έχει και μετά να εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα πιο διαφανές και πιο λειτουργικό πλαίσιο. Τέλος, αυτά είχα να πω γενικά και Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω. Αν κάτι αμέλησα και το ξέχασα να μου το υπενθυμίσετε να, το συζητήσουμε. Ολοκληρώνω και πάλι. Είμαι ευγνώμων για όλες τις παρεμβάσεις σας και προσβλέπω στη συνέχιση της εργασίας μαζί σας. Είναι μεγάλη αυτή η πρόκληση για μένα και με ιδιαίτερη χαρά εκδίωμαι σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Uh, well, <laughs> thank you. Ευχαριστώ, πάρα... Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κανιέτη και ζητώ συγγνώμη για την ε, παράληψη της ε, Λετωνίας. Βεβαίως για να υπερασπιστώ ότι... των Λετωνικών, με συγχωρείτε, για να υπερασπιστώ την γραμματεία μας προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε τη γλώσσα σας και ελπίζω σε επόμενη συνεδρία να μπορέσετε να μιλήσετε λετωνικά. Ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να επανέλθω στο γενικό ερώτημα για τα χρονοδιάγραμματα για τις εκθέσεις και την διαδικασία από εδώ και μπρος και τον συντονισμό για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή συνεδρίαση στο τέλος για να συντονιστούμε. Αυτό προτείνω. Οπότε θα ήθελα να περάσουμε... Ναι, ναι, όλα αυτά θα γίνουν στο τέλος. Αυτό είναι το καλύτερο νομίζω. Αλλά πρώτα απ' όλα θα έλεγα πως ε, οι εκθέσεις αυτές του συντονισμού είναι κάτι το πολύ σημαντικό όπως βλέπετε και οι συγητές συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και βέβαια στο να βρούμε τις προτεραιότητες θα είναι το πιο δύσκολο αλλά νομίζω πως ήδη συζητήσαμε και το έχουμε πει όταν έχουμε 50 προτεραιότητες δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα και η Κομισιόν θέλει να κάνουμε κάποιες πολιτικές επιλογές και ίσως χρειαστεί να ψηφίσουμε στο τέλος γιατί θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά παρόλα αυτά το συνολικό περιεχόμενο και η αξία που θα προσθέσουμε στις ε, προτάσεις Κομισιόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ανεξαρτήτω του ποιες προτεραιότητες θα δοθούν. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να περάσουμε να ακούσουμε συνεισφορές στην έκθεση Κορέα Ντεκάμπος. Να σου πω ποιου έχουμε στον κατάλογο των ομιλητών από πλευρά σκιωδών που είναι εδώ. Uh, Mrs. Uh, και εγώ είμαι επίση και ο δισηγητής, οπότε θα μιλήσω και εγώ λίγο. Ναι, ναι. Είστε, είστε. Πρέπει να μιλήσω πρώτος παρά το γεγονός ότι δεν είναι η σειρά μου, γιατί σε λίγο πρέπει να φύγω σε μια συνάντηση που έχει σχέση με τη Μέση Ανατολή και τα γεγονότα. Αν μου επιτρέπετε να πάρω τον λόγο. Right και ζητώ συγγνώμη από τους ε, συναδέλφους, αλλά επειδή οι δύο σκιώδεις εισηγητές από την ομάδα μου για τις άλλες δύο εκθέσεις δεν είναι εδώ, να μου επιτρέψετε να κάνω κάποια γενικά σχόλια που είναι οι θέσεις της ε, ομάδας που εκπροσωπώ. Το έγγραφο της Επιτροπής πολύ φοβούμαστε ότι ακολουθεί την ε, λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας η οποία σύμφωνα και με επίσημες τοποθετήσεις από την Κομισιόν δεν έχει εκπληρώσει τους στόχους της. Εμείς πιστεύουμε ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το όραμα της και να επανακαθορίσει τις προτεραιότητες της τόσο σε λεκτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο έτσι που να είναι αρκετά ορατή στους πολίτες. Η αγορά είναι χρήσιμη, έχει μάλιστα και τις αρετές της, δεν αποτελεί όμως αυτή καθεαυτή κοινωνικό μοντέλο. Η κοινωνική διάσταση πρέπει να καθιερωθεί ως η πρώτη προτεραιότητα και η νέα ατζέντα για την ενιαία αγορά πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτελεί και την πεμπτουσία της έκθεσης του κυρίου Ντεκάμπος, τον οποίον ευχαριστώ πάρα πολύ και μας βρίσκει συνοδοιπόρους σε αυτό το μονοπάτι. Ακόμη και σε μια κοινωνία ελεύθερης αγοράς δεν μπορούν τα πάντα να είναι προσπόληση. Δημόσια αγαθά και ανάγκες όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η κοινωνική ευημερία και η υγεία, η παροχή καθαρού πόσιμου νερού, ενέργειας δεν μπορούν να εξαρτώνται από δυνάμεις της αγοράς. Αυτό θα σήμαινε διάβρωση του ίδιου του συστήματος των εξουσιών όπως το καθορίζει η δημοκρατία. Ταυτόχρονα θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε δεν μπορούν να αγνοούνται. Εμείς πιστεύουμε ότι η προστασία του καταναλωτή και των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαμόρφωση αυτής της νομοθεσίας θα απαιτεί από τους νομοθέτες να υιοθετήσουν ένα νέο τρόπο σκέψης, να τοποθετηθεί η προστασία των καταναλωτών και η κοινωνική διάσταση ως μέρος του μηχανισμού ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη δημιουργία των νόμων και των κανόνων που υπαγορεύουν την ενιαία αγορά. Περαιτέρω, κάθε νομοθεσία που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη του αντίκτυπου της για την απασχόληση στον αντίστοιχο τομέα. Τονίζουμε ξανά ότι οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια ή γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο δεν πρέπει να καλύπτονται από το δίκαιο περί ανταγωνιστικότητα την νομοθεσία της ενιαίας αγοράς ή τους κανόνες για τη ρύθμιση των επιδοτήσεων ή την απελευθέρωση των δημόσιων συμβάσεων. Η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποτελεί κέριο πολιτικό ζήτημα. Τα καλά σχολεία και νοσοκομεία, το καθαρό νερό, οι ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές και η ενέργεια, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται στους περισσότερους ορισμούς μιας καλής ποιότητας ζωής. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω για μια συνάντηση που έχει σχέση με τα γεγονότα που τρέχουν στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυριάκο, για τη συνεισφορά σου και είμαι σίγουρος πως θα καταθέσει η ομάδα σου και οι τρεις όδεις ε, κάποιες τροπολογίες γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί η άποψη όλων. Οπότε, το δώσω τον λόγο στην κυρία Τούν για να παρέμβει και εκείνη αν είναι έτοιμη. Να έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σκιώδης ε, συγκεντρία το δεύτερο κομμάτι του κυρίου Κορέρα Ντεκάμπο. Είχαμε μια συνεδρίαση ε, πολύ επικοδομητική τη Δευτέρα που μα πέρασε συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία, αλλά βεβαίως έμειναν ανοιχτά. Θα έλεγα πως η γενική μου στάση είναι πως δεν θα πρέπει να μην αντιδράσουμε σε αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν, αλλά όπως είπε και η κυρία Κανιέτα, χρειαζόμαστε μια ενεργή προσέγγιση με σαφείς προτεραιότητες, προτάσεις και κατάταξη αυτών των προτεραιοτήτων. Επίσης έχω ένα πρόβλημα και στα πολωνικά με τη μετάφραση της λέξης διακυβέρνηση. Πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα, μια κοινή προσπάθεια και πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές στη γλώσσα μας. ορίζω το ότι συμφωνούν στην ίδια δομή οι εισηγητέ και στις τρει εκθέσει, οπότε δεν ξέρω ποια θα είναι η τελευταία πρόταση του κυρίου Κορέρα Ντεκάμπος, γιατί υποθέτω πως θα έχει την ίδια μορφή με τις άλλες εκθέσει. Αυτό το οποίο είδα εγώ μέχρι τώρα. Έχω πολλές παρατηρήσεις εκεί πέρα, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τη δομή της έκθεσης. δεν αναφέρονται οι, ξεκάθαρα οι προτεραιότητές μας και δεν υπάρχει οργάνωση στην ιεραρχία αυτή που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Απαριθμοί, πρωτοβουλίες που περιέχονται στην νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς αλλά δεν δείχνει σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Και από ό,τι κατάλαβα η δομή θα αλλάξει είναι διαφορετική η δομή από αυτά τα οποία ακούω από τους άλλους, από τις άλλες δύο εκθέσεις. Όσον αφορά δε το περιεχόμενο, δεν είμαι σίγουρη για το εάν χρειαζόμαστε τρεις ε, σελίδες προθέσεων, γιατί είναι δύσκολα. Δύσκολο να το διαβάσει κανείς. Συμφωνήσαμε πως ε, θα καταλήξουμε σε μια διακομματική προσέγγιση Έχουμε λοιπόν κάποια σημαντικά επίμαχα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η διάσημη εισαγωγή οριζόντιας κοινωνικής ρήτρα, όπου δεν αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα μετρηθεί και πώς θα λειτουργήσει. Οπότε νομίζω πως πρέπει να πάμε προς την κατεύθυνση Τη διακομματικής προσέγγιση για να καταλήξουμε κάποτε σε ένα καλό έγγραφο. Η έκθεση του δεύτερου μέρους έχει επίσης ε, σημαντικό κεφάλαιο 3 που λέγεται κενά, χάσματα. Όπου δεν νομίζω πως πρέπει να επικεντρωθούμε στα κενά, αλλά να κάνουμε σαφείς προτάσεις. Και η έκθεση δεν ε, δίνει βάρος στο δεύτερο μέρος. Κάποια από αυτά τα χάσματα που λέτε αντιμετωπίζονται από άλλα σημεία του νόμου περί εσωτερικής αγοράς, ειδικά το, το πρώτο μέρος, όπως ε, πνευματικά δικαιώματα, ψηφιακή ενιαία αγορά, το ίδιο. Και για αυτό το οποίο λέτε βραχυπρόθεσμες προτάσεις, που εγώ θεωρώ πως πρέπει να ονομάσουμε προτεραιότητες, όπως πειρατεία, κλεψίτυπα προϊόντα. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία με άλλους ηγητές. Επίσης, πολιτική επικοινωνία. Συμφωνώ με την κυρία Ρούλε πως ε, η διαδικασία της, της ε, διαβούλευσης δεν λειτουργεί. Θεωρώ πως εδώ πέρα πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα με τους ηγητές στο μέρος 3 και να μην τα γιατί δημιουργείται σύγχυση. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ιεραρχία και σαφεί προτεραιότητες, το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να είναι αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, ασφάλεια προϊόντων, διεπιτήρηση δηλαδή της αγοράς, φάσμα, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, αν είναι 5 με 7 οι προτεραιότητε, νομοθετική πρόσβαση σε συγκεκριμένε. Ε, τραπεζικές υπηρεσίες. Επίσης από τις προτάσεις Κομισιόν νεολαία κινήσει, αυτοκίνητα και, εάν μου επιτρέπετε, περιαγωγή δεδομένων και φωνής και ενιαία αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, και σκέφτομαι εδώ πέρα τα πακέτα, τα δέματα. Ο κύριος Μπούσα το έχει αναφέρει και στην έκθεσή του και βεβαίως μετά θα έχουμε έτσι μια πιο σαφή έκθεση. Τους θα έχει μεγαλύτερη συνοχή με αυτά τα οποία λένε οι άλλοι εισηγητές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Τούν. Τώρα, Κρόιτσμαν και η κυρία Ρίλε. Και η κυρία Γκέπχαρτ νομίζω θέλει να παρέμβει. Θα μιλήσετε λοιπόν μετά τους σκιώδησίτες. Κάποιος άλλος ε, θέλει να λάβει τον λόγο. Ναι, οπότε, Κρόιτσμαν και μετά Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κορέα Ντεκάμπος για τη δουλειά που έκανε, αλλά να κάνω και μια σειρά προτάσεις και βελτίωση. Πρώτα απ' όλα η δομή. Καλύτερο θα ήταν η έκθεση αυτή να ε, οργανωθεί αναθέματα όπως και οι άλλες εκθέσεις για την, για την ομοθεσία περί ιστορικής αγοράς. Οι τίτλοι της αιτιολόγησης αναφέρω κοινωνικά δικαιώματα, δικαιώματα καταναλωτών, ελεύθερη διακίνηση θα μπορούσαν να αποτελέσουν βεβαίως ε, κάποιο υπόδειγμα και θα πρέπει να δούμε καλύτερα τις προτεραιότητες για να δώσουμε περισσότερες, ένα προσανατολισμό στην Κομισιόν για την ουσία συμφωνώ πως η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ε, στον τομέα ενέργεια και ψηφιακή οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική στόχη για την ολοκλήρωση αυτής της αγοράς, ε, κάτι το οποίο θα έχει αυτά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε δεν χρειαζόμαστε οριζόντια κοινωνική ρήτρα, είπε η συνάδελφος, η οποία θα πηγαίνει πέρα από τις υπάρχουσες διατάξεις. Ήδη η νομοθετική πρόταση της, οι νομοθετικές προτάσεις Κομισιόν θα εξετάζονται ως προς τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Οπότε σημαίνει πως θα συμφωνούν οι νόμοι με την ε, συνθήκη, το άρθρο 9 και με την χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την δε οδηγία περί θα πρέπει να ξεχαρίσουμε πως δεν χρειάζεται αλλαγή της υπάρξεως οδηγίας. Αντιθέτως, Κομισιόν και κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν, να ξεκαθαρίσουν σημαία τα οποία εμποδίζουν την ενιαία και απρόσκοπτη εφαρμογή. Επιπλέον, δεν χρειαζόμαστε μία οδηγία πλαίσιο για τις ε, γενικότερες ε, για το Γενικό Δίκαιο των ε, Δημοσίων Προμηθειών, καθώς υπάρχουν ήδη σχετικές οδηγίες και βεβαίως αν εφαρμόζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν σημαίνει πως είναι υποχρεωτικά με αρνητικές κοινωνικές ε, συνέπειες. Υπάρχει η δυνατότητα στους διαγωνισμούς, της δημόσιας προτιμήθειες να υπάρχουν ειδικέ τομεακές απαιτήσει. Ακόμα και ο Μάριο Μόντι στην έκθεσή του, στην έκθεση επιτροπής του, είπε πως δεν θα πρέπει να πάμε προς αυτή η κατεύθυνση καθώς γίνονται μετά πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες ε, για ενιαία αγορά Επίσης, ε, αναλόγες διαδικασίες θα πρέπει να περιοριστούν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δικαϊκά στήματα τα οποία υπάρχουν, για να μην οδηγηθούμε σε μαζικές αγωγές σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο. Συγκεκριμένα μετά δύο προτάσεις της Κομισιόν είναι πάρα πολύ υποσχόμενες. Η εισαγωγή επαγγελματικής ταυτότητας για καλύτερη κινητικότητα των ε, εργαζομένων καθώς και η καλύτερη πολιτική όσον αφορά το ευρυζωνικό ίντερνετ και την πολιτική του φάσματος. Η κυρία Ρούλη. Για τα, αυτά τα τελευταία σημεία συμφωνώ με τον κύριο Κρόισμαν. Πιστεύω ότι σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση θα διευκολυνόμαστε αν είχαμε την αμοιβαία αναγνώριση και αυτό θα έπρεπε να εγγραφεί ως σημείο και κατά τα ε, άλλα για τα το ευρυζωνικό φάσμα και το roaming την περιαγωγή και τις ε, διασυνοριακές ε, διαβιβάσεις δεδομένων πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό. Είναι λίγο εξειδικεύει το θέμα αυτό, πολύ λίγο κύριος Κορέα. Όμως κατά τα άλλα το βρίσκω σωστό ότι την οδηγία περί αποστολής, περί απόσπασης εργαζομένων πρέπει να μας κάνει να έχουμε μια επικαιροποίηση και προσαρμογή. Γνωρίζετε ότι κύριε Κρόσμαν εμείς ε, είχαμε υποστεί επιπτώσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ε, νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά συναφή απόφαση και όσον αφορά και τις, τα δικαιώματα αμοιβή μισθολογικά αλλά και για την οδηγία περί απόσπασης. Είναι ένα γερμανικό πρόβλημα όμως παραμένει ευρωπαϊκό πρόβλημα ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση στην οποία πρέπει να καταλήξουμε και μια εξειδίκευση ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια Διαφωνώ λοιπόν σε σχέση με αυτό μαζί σας. Και όσον αφορά και την ε, ένταξη ή ε, κατακύρωση, είχαμε εργαστεί για αυτό το θέμα και είχαμε προβλήματα με την κοινωνική υπεύθυνη πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση. Έχει και ε, μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπεται σχετικά. Το χαιρετίζουμε αυτό. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνιση. Τι είναι αποσαφήνιση, τι είναι δυνατόν να γίνεται και τι όχι. Και σε σχέση και με τα περιβαλλοντικά κριτήρια κριτήρια και σε σχέση και με τα κοινωνικά κριτήρια κάτι τέτοιο που δεν γίνεται πρέπει για αυτή την οδηγία να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Δεν θέλω να πάω ιδιαίτερα σε λεπτομέρειες αλλά αυτό το πεδίο αντί να μιλάμε όλο για ένα πλαίσιο πρέπει πιο εξειδικευμένα να δούμε αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αποσαφινιστούν για να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά και την παροχή υπηρεσιών γενικού ε, συνολικού συμφέροντος. Και έχει προαναγγελθεί ότι το πλαίσιο ενισχύσεων επιδοτήσεων θα επανεξεταστεί και το θέμα της κατακύρωσης. Αυτά τα δύο πρέπει να αποσαφινιστούν, είναι σημαντικά. Ζήτησα όμως τον λόγο να παρεμβώ, διότι κάποια σημεία σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Κορέα τα βρίσκω προβληματικά. Δίνει συνέχεια στην πρόταση της Επιτροπής ο κύριος Κορέα όσον αφορά τα δάνεια από τα ενυπόθηκα δάνεια. Είναι όμως ε, πολύ, πολύ μικρή εξειδίκευση. Όταν γίνεται λόγος για αυτό το θέμα και αναφέρομαι στο αγγλικό παράθεμα, άμεση δράση για μια ενιαία αγορά ενυπόθηκων δανείων, θα πρέπει εδώ να δούμε ότι αυτά τα δάνεια ήταν κίνητρο ε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που οδήγησε ως αίτιο σε κρίση. Αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα εναρμονισμό, πρέπει πρώτα να αποσαφινιστεί Πώς θα υπάρξει ένας τέτοιος εναρμονισμός χωρίς να υπάρξει επιβλαβής επίπτωση στις αγορές. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι προβληματικό να ζητήσουμε να υπάρξει έτσι συλλήβδη εναρμονισμός. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί η προστασία καταναλωτών σε αυτό το πλαίσιο. Και η διαφάνεια είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Εδώ όμως βιαστικά και συλλήβδην να ζητάμε να εναρμονιστεί ο τομέας των ενυπόθηκων δανείων είναι προβληματικό. Να συζητήσουμε πρώτα παρακαλώ σε βάθος προτού υπάρξει ε, μήνυμα που θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συμφωνούμε με ένα τέτοιο εναρμονισμό διότι δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίπτωση ενός τέτοιου μέτρου. Θέλω και άλλα να αναφέρω, αλλά σε σχέση με την πρόταση Μπαρνιέ θεωρώ ότι υπάρχουν ελλείψεις. Είναι το θέμα της αντιμετώπισης των κλιματικών ε, φαινομένων και της ε, ε, μεταβολής της κλιματικής, των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει εδώ να το τονίσουμε αυτό περισσότερο όσον αφορά την αηφορία της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Ρούλε. Κάποιες παρατηρήσεις ως σκιώδης για την έκθεση αυτή θα κάνω τώρα. Πρώτον, κατανοώ κάποιες από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων του κ. Κρότσμαν και της κ. Ρούλε ιδίω. Συμφωνώ με την κυρία Ρούλε κυρίω για το ότι η ενιαία αγορά υποθηκών, υπονυπόθηκων δανείων είναι σημαντική. Ιδίω για την ανάγκη της υπεύθυ, του υπεύθυνου δανεισμού και των σχετικών μέτρων Ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα υπάρξει πραγματική διασυνορική αγορά στεγαστικών δανείων που περιλαμβάνουν πολλούς κινδύνους. Πάντως έχω την εντύπωση ότι πιο ενδεδειγμένο ίσως για τα συμφέροντά μας θα ήταν να ζητήσουμε από την Επιτροπή να κάνει μία έκθεση για την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την καταναλωτική πίστη σε ό,τι αφορά την, ε, που είναι σημαντικότεροι για τη συμμετοχή των πολιτών στην ενιαία αγορά. Επίση, για πρώτη φορά είδαμε στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη ρυθμίσει για την ανάγκη υπεύθυνου δανεισμού, καλύτερη ενημέρωσης που ισχύουν για όλη την Ένωση. Και αυτό είναι σημαντικό δεδομένων των τεράστιων αποκλήσεων στο ποσοστό χρήσης ε, της πίστης στην ενιαία αγορά και αυτό είναι πιο σημαντικό για μας. Ίσως λοιπόν να προτείνω κάποιες τοπολογίες σχετικά. Δεύτερον, το θέμα των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, γενικού συμφέροντο. Η οδηγία, αυτό το ζήτημα εμφανίζεται συνεχώ τα τελευταία 11 χρόνια που είμαι στο Κοινοβούλιο. Και πάντα το ίδιο πράγμα από αυτούς που υποστήριζουν την ιδέα αυτή. Δεν καταλαβαίνω τα προβλήματα που θέλει να λύσει η οδηγία αυτή. Είπα και νωρίτερα ότι η, τούτο αποτελεί μια λύση που αναζητεί πρόβλημα. Δεδομένου του ότι θα έχουμε μια μεγάλη αναθεώρηση των ε, διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων σε κάθε περίπτωση και η Επιτροπή έχει ζητήσει μια σειρά, να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων, παροχές, ε, εκχώρηση υπηρεσίας, ε, τι θέλουν να κάνουν οι αρχές, μια σειρά νέων κλάδων αλλά και τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Μια απόφαση για το, την οδηγία πλαίσιο που είπα παραμένει ασαφέστατη. Καλύτερα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί μπορούμε να κάνουμε πολιτική πρόοδο. Διότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι τα κρατη μελε ενδιαφέρονται για μια, αυτή την ε, μυθική οδηγία πλαίσιο. Μπορεί οι άλλοι συνάδελφοι βέβαια να θέλουν να διαφοροποιηθούν, αλλά εγώ πάντως αυτή τη θέση έχω. Δύο παρατηρήσεις ακόμα. Ένα από τα θέματα που έθεσε η Επιτροπή στον κύριο Μπαρνιέ, δεν ξέρω το θυμάστε, και είχε προχωρήσει σε κάποια σχόλια, αφορούσε το γεγονός ότι η εικόνα της ενιαίας αγοράς στους πολίτες χρωματίζεται από το ότι οι κινούμενοι οι πολίτες ε, στην Ένωση θεωρούν ότι τα δικαιώματα που θεωρητικά πρέπει να έχουν απλή τρόπη μεταφοράς, δικαίωμα να μετακινήσουν ε, την οικογένειά του από χώρα σε χώρα, να ανοίξουν ένα λογαριασμό, να αλλάξουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων, να μεταφέρουν τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα, να τα βρουν με τις φορολογικές υπηρεσίε, να, πέρα, να πάνε τα παιδιά του στο σχολείο με απλή μεταφορά των επαγγελματικών εκπαιδευτικών ε, προσόντων, δεν γίνονται από τα κράτη-μέλη. Απλώς και μόνο. Είδατε την έκθεση του κυρίου Λαμασούρ που ανέλαβε η κυρία Ρέντινγκ σε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για τους πολίτες στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Είναι απογοητευτικό το ότι δεν υπάρχει μεγάλη παραπομπή στην την έκθεση αυτή και το ότι ο κύριος Μπαρνιέ μας είπε ε, ότι θα έρθει, ε, θα μας φέρει έναν κατάλογο με τις βασικές ενοχλήσεις, τις 20 βασικότερες ενοχλήσεις της ενιαίας αγοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη. Εμείς δεν απαντήσαμε επίσημα στην έκθεση Rending, διότι δεν ε, μπορούσαμε λόγω του ότι είχαμε το νομοθετικό κείμενο για την ενιαία αγορά, αλλά με απογοήτευσε το ότι κανία, καμία άλλη Επιτροπή στο Κοινοβούλιο δεν θεώρησε ότι θα μπορούσε να αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή και να κάνει μια έκθεση. Γιατί στο τέλος τέλος εδώ είμαστε για να εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και την ενόχληση των πολιτών. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να γίνει μια σχετική μνήα. Ένα ακόμα στοιχείο που μπορεί να θέλουμε να παρουσιάσουμε στην έκθεση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δεκάμπος θέλει να κάνει μια, ένα τέτοιο σχετικό σχόλιο. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη σπουδαιότητα της μεταρρύθμισης της πρότασης για την αμοιβαία αναγνώριση. Να την αναδείξουμε. Κάποια θέματα, όπως επαγγελματικές κάρτες, είναι σημαντικό. Αλλά μια επαγγελματική κάρτα είναι σημαντική μόνο για τις πληροφορίες που περιέχει θα μπούμε όμως και σε επικίνδυνα ζητήματα, φερρυπίν, κατά ε, ε χρησιμοποίηση από κοινού στοιχείων ε, μεταξύ επαγγελματιών, ιατρικών στοιχείων ενδεχόμενα. Θα δούμε ζητήματα όπως την μεταφορά και χρήση των προσωπικών δεδομένων. Μια διάσταση κατά άποψή μου σημαντική. Εκεί τα συμφέροντα των πολιτών και τα συμφέροντα της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να συμφιλειωθούν πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι νομίζω ότι προσεγγίζουν το ένα το άλλο. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι το θέμα των τραπεζικών υπηρεσιών, ε, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και άλλες διαστάσεις είναι σημαντική προτεραιότητα γιατί και αυτές επηρεάζουν σχεδόν όλους τους πολίτες. Και κλείνω με ένα βασικό ζήτημα κατά την άποψή μου. Η κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς και ο κοινωνικό τη αντίκτυπο. Όταν βλέπουμε αυτή τη διάσταση θα πρέπει να δώσουμε την κύρια πρωταρχική έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Και δεν περνάει αυτό επαρκώς εμφανώς στην έκθεση. Αν δεν δημιουργήσει με επιτυχία νέες θέσει εργασία η ενιαία αγορά, μακροπρόθεσμε θέσει εργασία με προοπτικές, ιδίως στις νέες επενδύσεις, θα έχουμε αποτύχει στις προσδοκίες των πολιτών. Και ο κοινωνικός αντίκτυπος μιας αγοράς που δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας θα είναι εξαιρετικά βαθύς με τεράστιες επιπτώσεις. Θα έπρεπε λοιπόν να συνδέσουμε τα ζητήματα αυτά, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ο αντίκτυπο της αλλού στις επιχειρήσεις, στη χρηματοοικονομική αγορά θα ήταν θετικό. Αλλά νομίζω ότι η αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει σαφέστερα την ανάγκη να δημιουργούνται θέσεις εργασία για να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτά ήθελα να σας πω. Μίλησα ε, με τον κύριο Ντεκάμπος για τα ζητήματα αυτά και περιμένω τις, ε, τα σχόλιά σας. Τρεις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο τώρα. Έχουμε χρόνο συνάδελφοι για όλες τις εκθέσεις. Γκέπχαρτ Βάιλερ Μάγερ. Κανείς άλλος. Κατόπιν η Επιτροπή θα μιλήσει και ο κύριος Δεκάμπος κατόπιν. Κύριε Γκέπχαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Κορέντε Κάμπος για την πραγματικά πολύ καλή και σε θέματα αρχών συνεργασία. Και θα ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό το τμήμα της πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εκείνο που τις μεγαλύτερες σε βάθος ε, ε, αλλαγές χρειάζεται διότι αυτό αποτελεί τον πυρήνα την πεμπτουσία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι ο τίτλος ήδη της πρότασης Μπαρνιέ είναι η ενιαία εσωτερική αγορά αηφορία πώς θα αναφέρεται ανταγωνιστική ενιαία εσωτερική αγορά. Ξέχασα τον τίτλο, συγγνώμη, για τους πολίτες, έτσι για τους πολίτες. Υπό το πρίσμα ότι οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Για αυτούς τους λόγους είναι σε αυτό τον τομέα αναγκαίο να δούμε αυτή την προσέγγιση σε βάθος. Μετά ο κ. Κορέντε Κάμπος τι κάνει έχει ουσιώδης έργο που αναπτύσσει και θα έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια απάντηση σε αυτά που η κυρία Κανιέτε καθότι γνωρίζω ανέφερε. Μια κοινή συνιστόσα και στις τρεις κοινέ εκθέσεις. Δηλαδή επί της ουσίας τοποθετήσεις πώς αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως γίνεται από την έκθεση Κορέα Ντεκάμπος με μια κοινή προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί όσον αφορά την κοινωνική ρήτρα, κοινωνικές διατάξεις, την υλοποίηση εκείνων που είναι καινούρια στοιχεία στη συνθήκη της αγοράς, δηλαδή την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το άρθρο 9 αναγνώρισε ότι υπάρχουν υπηρεσίες καθολικού συμφέροντος προς ε, το ε, ολικό συμφέρον και της χάρτας των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά να αποτελέσουν μια κοινή βάση. Κοινά θεμέλια, κοινή συνιστόσα και στι τρει εκθέσει. Καλή υπόθεση, καλό θα ήταν αυτό. Εκείνο όμω στη συνέχεια που συνέβη με τον κύριο Κορέα Ντεκάμπο, επειδή υπήρχε μικρό χώρο ε, γι' αυτό, ήταν το πέμπτο τμήμα δεν εντάχθηκε. Ε, και γι' αυτό, Αντώνιο, θα πρέπει το πέμπτο τμήμα να, ε, να ενταχθεί με τροπολογίε που θα θέτουν τι προτεραιότητε. Ε, διαφορετικά μέλη, διάφορα μέλη έθιξαν αυτέ τι προτεραιότητε και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε ώστε να ενταχθεί αυτό το τμήμα στην έκθεση. Αυτό πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Σε δύο σημεία θα ήθελα να διαφωνήσω με τον πρόεδρο Μάκομ Χάμπορ. Ποια είναι αυτά τα δύο σημεία. Δύο σημεία. Διαφωνώ δυστυχώς μαζί σας κύριε Χάμπορ. Πρώτον, ο κύριος Κορέντε Κάμπος ήθελε τις προτάσεις της κυρίας Ρέντινγκ να τις ε, εντάξει και να τις ε, ε, συνεκφωνήσει. Εγώ στην τελευταία συνάντηση συντονιστών πρότεινα να το κάνουμε αυτό. Οι άλλοι όμως συντονιστές το απέρριψαν. Και γι' αυτό ο κύριο Κορέντε Κάμπος δεν μπόρεσε να εντάξει αυτό το στοιχείο. Δεν υπήρχε πλειοψηφία από πλευρά τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή να πούμε ναι, πρέπει να προλιανθεί το έδαφο με αυτέ τι προτάσει τη κυρία Ρέντινγκ. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον κύριο Κορέντε Κάμπο για το ότι δεν το έκανε δεν επιτρεπόταν να το κάνει και έτσι τήρησε την απόφαση που είχαμε λάβει, πράγμα το οποίο με κάνει να λυπούμε για αυτή την κατάσταση. Θλίβομαι γι' αυτό. Αν ο πρόεδρο και οι άλλοι είχαν διαφορετική άποψη, ευχαρίστω ο κύριο Κορέντι Κάμπο θα είχε εντάξει αυτό το σημείο. Τώρα πρέπει με τροπολογίε να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε και να δούμε ποια θα είναι η τοποθέτηση τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή στο τέλο. Το δεύτερο στο οποίο διαφωνώ μαζί σα, κύριε Πρόεδρε Μάκομ Χάρμπορ, είναι το ότι όταν λέτε ότι χρειάζεται μια ρύθμιση για την ε, ε, διάταξη υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος. Είπατε ότι είναι μια λύση η οποία αναζητεί το πρόβλημά της. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Πρώτον, δεν είπαμε ότι θέλουμε μια οδηγία πλαίσιο, αλλά ότι θέλουμε ένα νόμικο πλαίσιο. Αυτό είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Δεν καθορίζεται πώς αυτό θα γίνει. Αυτό θα αποτελέσει θεμέλιο για τη συζήτηση του μέλλοντος. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε σε αυτό, σε, αυτό τον τομέα και τι θέλουμε να κάνουμε. Χρειάζεται μια κοινή γραμμή πλεύσης ε, από το Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία δεν καταλήξαμε ακόμα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καθορίσουμε ότι θα είναι μια οδηγία, ένα κανονισμό ή οτιδήποτε. Ζητούμε όμω ένα νομικό πλαίσιο να εισαχθεί. Δεύτερον, στη συζήτηση για την οδηγία περί παροχή υπηρεσιών το είδαμε αυτό σε σχέση με συζητήσει που διεξήχθησαν όταν είχαμε το πεδίο εφαρμογή για αυτή την οδηγία περί παροχή υπηρεσιών. Αν θα είναι υπηρεσίε στην υγεία, κοινωνικέ υπηρεσίε και για άλλου τομεί που ουσιώδη σημασία, σπουδαιότητα έχουν για του πολίτε. Αν θα είναι εμπορευματοποιημένες τέτοιες υπηρεσίες ή όχι εμπορικού χαρακτήρα ή κερδοφόρου χαρακτήρα. Και είπαμε όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Χρειάζονται ειδικέ διατάξει και εξειδίκευση για όλα αυτά τα θέματα που θα ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Διότι για του πολίτε στον τομέα τη υγεία οι πολίτε δεν είναι καταναλωτέ αλλά ασθενεί. Και οι ασθενεί έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα προστασία και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη σύνδρομη και δεν είναι καταναλωτέ που αγοράζουν κάτι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εδώ μια διαφορετική προσέγγιση, διαφοροποιημένη προσέγγιση. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω στον κύριο Κρότσμαν ότι πρέπει να διαφωνήσω δυστυχώς μαζί του. Γι' αυτό, σε σχέση με την κοινωνική ρήτρα, το ότι αυτό ήδη γίνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπούμε γι' αυτό. όμως. Κοινωνικέ αποτιμήσει ή αξιολογήσει δεν γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάξει μόνο οικονομικέ ε, επιπτώσει ε, αναλύονται και εξετάζονται γι' αυτό εμεί οι σοσιαλδημοκράτε θεωρούμε ότι μια κοινωνική ρήτρα συνεισφέρει πολύ περισσότερο και δεν βλέπει μόνο οικονομικέ επιπτώσει που αξιολογούνται αλλά πολύ περισσότερο τα κοινωνικά θέματα εντάσσει οι κοινωνικέ επιπτώσει τη νομοθεσία στα δικαιώματα των πολιτών ήδη κατά την ε, δημιουργία ενός νομικού πλαισίου πρέπει να συνεξετάζονται ως θέματα. Και έτσι και να μην κάνουμε αυτό το οποίο προβλέπετε τώρα, τι θα ποιες, τι θα συνεπαγόταν αυτό οικονομικά. Πολύ πιο πριν πρέπει να εντάξουμε στην νομοθετική μας προσέγγιση τα κοινωνικά θέματα, με την κοινωνική ρήτρα, πώς αυτά θα διαμορφωθούν και να, συμπ, να προβληματιστούμε όχι ποιε θα είναι οι επιπτώσεις μόνο στην οικονομία, όχι μόνο ποιε θα είναι οι επιπτώσεις στην ενιαία εσωτερική αγορά, αλλά να προβληματιστούμε τι θα σημαίνουν όλα αυτά για τους πολίτες, για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, για τα, ποιες επιπτώσεις θα έχει στους πολίτες ως καταναλωτές και ποιε επιπτώσει θα έχει στου πολίτε ω εργαζόμενου συνολικά. Αυτή την ολιστική, συνολική προσέγγιση που και ο κύριο Γκρέκ είχε εντάξει στη δική του έκθεση. Αυτά είναι πολύ σπουδαία θα έλεγα εγώ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη διότι πρέπει να αποχωρήσω και εγώ, διότι για τον πίνακα, για την ψηφοφορία, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για αυτή την οδηγία που πρέπει να προετοιμάσω για το απόγευμα για την ομάδα μου. Υπάρχουν κάποια θέματα που εκκρεμούν και πρέπει να απαντηθούν και πρέπει εγώ να ε, συνεισφέρω σε αυτές τις απαντήσεις και πρέπει να αποχωρήσω. Όμως μια προσέγγιση προς τον κύριο Μπουσόη και την έκθεσή του θα ήθελα να κάνω. Παραμείνετε κύριε Μπουσόη και προσέξτε τι θέλω να πω γιατί κάποιες παρατηρήσεις ήθελα να κάνω προς εμάς. Ίσως όμως σας παρανόησα και εσάς και ε, σε σχέση με την απάντησή σας θα μου τη διαβιβάσουν ε, οι συνεργάτες μου γιατί δεν θα παρίσταμε όταν θα απαντήσατε. Μιλήσατε για τον τομέα της καινοτομίας, για το τι θα έπρεπε να γίνει. Έχετε δίκιο, σας δίνω δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει να μας προβληματίσει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η ερώτησή μου προς εμάς κύριε Μπουσόη είναι πώς θα θέλατε εσείς να το αντιμετωπίσετε αυτό. Διότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις αναμεταξύ τους. Ξέρω για παράδειγμα ότι η Γαλλία έχει το όραμα μιας ε, τέτοιας ε, μεγάλης κοιλάδας ε, σίλικων του πυρητίου στη Γαλλία για την τεχνολογία και τις επικοινωνίες και την πληροφορική. Εμείς στη Γερμανία εργαζόμαστε σε μικρότερο, μικρότερη κλίμα, κλίμακα όσον αφορά τις ε, ομάδες κατηγοριοποιημένα clusters ε, που συνεισφέρει στο να δημιουργηθούν τέτοιες ομάδες επιχειρήσεων ως θεμέλιο της καινοτομίας ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό προάγει περισσότερο. Αυτά εργαζόμαστε υπομορφή clusters, υπομορφή τέτοιων ας έλεγα τσαμπιών, βοστρίχων. Πώς θα μπορούσαμε να, ε, να καταλήξουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τι θα έπρεπε να γίνει. Θα ήθελα περισσότερο να ζητήσω να αποσαφηνίσετε τα πράγματα σε σχέση με την ε, ανάπτυξη και την αηφορία. Τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουμε, προστασία περιβάλλοντος, προστασία έναντι των κλιματικών αλλαγών, αυτά να ενταχθούν πολύ περισσότερο για την αηφορία και την ανάπτυξη. Αν θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό στην έκθεσή σας, καλό θα ήταν έτσι ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύλεν. Κάποια σημεία που απευθύνες προς εμένα. Είπα στην εισαγωγή μου πως θεωρώ πως ε, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στην έκθεση Reading που χρειάζεται άλλη μια έκθεση. Α, υπάρχει λόγος να κάνουμε παραπομπέ. εκεί πέρα. Αυτό έλεγα ε, σε σχέση με τις ε, τροπολογίες, γιατί ήθελα να μείνουμε στο πλαίσιο αυτό για την οδηγία πλαίσιο αυτό ανέφερε ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος. Οπότε θα συνεχιστεί η συζήτηση πάνω σε αυτό. Και αναμένω βεβαίως τον ορισμό του προβλήματος που λύνουμε εδώ πέρα, τον ορισμό σας. Και θα φροντίσω βεβαίως να ακούσει αυτά τα οποία είπατε ο κύριος Μπιζόη. Και τώρα η κυρία Βάιλερ και Μάιερ. κυρία Βάιλερ πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα μετά τη συζήτηση αυτή της έκθεσης και τις συνεισφορές των συναδέλφων από τις άλλες ομάδες να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κρότσμαν, ο οποίος ε, δεν ε, παρακολούθησε όλη τη συζήτηση για την οδηγία των υπηρεσιών. Να του συστήσω λοιπόν να δει την πρότασή μας για την πρόταση πλαίσιο για τις υπηρεσίες της κοινοφελής. Δεν ήταν ε, κάτι το οποίο κάναμε εύκολο και δεν θέλαμε βεβαίως να διαλύσουμε αν θέλετε το δίκαιο των διαγωνισμών των δημοσίων προμηθειών. Αντίθετο, θέλουμε να το συμπληρώσουμε όπω κάνει και ο Επίτροπο Μπαρνιέ, ο οποίο σκέφτεται μήπω θα μπορούσαν να γίνουν δεσμευτικέ ή κοινωνικέ ρήτρε. Νομίζω πως σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο τον Απρίλιο και τον ρωτήσαμε κάτι σχετικό στις Κροάσεις και μιλήσαμε και με δημάρχους για το αν θέλει να κάνει η Ευρώπη κάτι τέτοιο. Πρόκειται λοιπόν για μια μεταξέλιξη κάνουμε δηλαδή πιο συγκεκριμένα τα πράγματα μπορούν να γίνουν εκεί πέρα. Αυτός είναι ο στόχος, όχι να αλλάξει ή να αποδιοργανωθεί το δίκαιο των δημοσίων προμηθειών. Αυτό είναι λάθος. Δεύτερον, όταν λέτε πως οι κοινωνικές επιπτώσεις θα πρέπει καλύπτονται ήδη από τις ε, μελέτες επιπτώσεων. Να σας πω πως ε, πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες νομίζω εγκρίναμε την έκθεσή μου, τη γνωμοδότηση για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων που βεβαίως θα πάει μετά στην κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ψήφισε η Επιτροπή μας πως θα πρέπει να δούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις πιο πολύ στην αξιολόγηση επιπτώσεων από ότι τώρα αυτό συμβαίνει πως δεν λαμβάνει χώρα επαρκώς αυτή τη στιγμή και πρέπει η Κομισιό να το κάνει καλύτερα από ό,τι μέχρι στιγμής. Οπότε δεν καλύπτεται. Τέλος. Ε, η επαγγελματική αυτή ταυτότητα αναμένω με αγωνία και για τις 50 αυτές τις προτάσεις για το τι θα γίνει στην οδηγία γιατί πριν δούμε την ομοθεσία δεν μπορούμε να κρίνουμε τι μορφή θα έχει. Εγώ έζησα και τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, για την ταυτότητα κινητικότητα των νέων και αναρωτιέμαι τι απέγινε αυτή. Το είχαμε εγκρίνει με μεγάλο ενθουσιασμό, νομίζω η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων επίσης μαζί μας και διαπιστώνω πως πάρα πολλοί νέοι που τελειώνουν ε, το σχολείο και το πανεπιστήμιο δεν ξέρουν καν για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν τι είναι αυτή η ταυτότητα κινητικότητα. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί για να τους δώσουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουν και κάποια συν για τους ε, εργοδότες. Και δεν έχει νόημα βεβαίως αν δεν συμμετέχουν και οι εργοδότες, γιατί θα πρέπει να δεχτούν αυτοί αν θέλετε αυτές τις ταυτότητες και να αναγνωρίσουν ε, τους πόντους ή τα πιστοποιητικά που θα περιέχονται εκεί μέσα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους αξιολόγηση επιπτώσεων για να δούμε τι έγινε από τα πιστοποιητικά αυτά κινητικότητας για τους νέους πριν κάνουμε το ίδιο πράγμα για τους ενήλικους και τους λοιπούς εργαζόμενους. Μην κάνουμε δηλαδή πάλι το ίδιο λάθος, να δημιουργήσουμε μεγάλες προσδοκίες, θα έχουν όλοι αυτά τα ωραία μπλε τις μπλε ταυτότητούλες. Αυτό δηλαδή με, με τους νέους έχει γίνει τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια, 7-8 χρόνια. Οπότε πολλά πράγματα επαναλαμβάνουμε στα 50 αυτά σημεία. Θα ήθελα να γνωρίσω λοιπόν τι απέγινε αυτό, τι πήγε τότε στραβά, γιατί μόνο εάν το ξέρουμε μπορούμε να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Ωραία, ευχαριστώ. Μπορούμε να, να τα δούμε αυτά. Είναι, είναι σωστά πράγματα και μπορείτε να τα συζητήσετε με τον εισηγητή. Κυρία Ρούλε, νομίζω... Ναι, και, και στην πρώτα 34 συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο. Οπότε ίσως θα πρέπει να ενισχυθεί εκεί η πρώτα 34. Ο κύριος Μάιρ τώρα, τελευταίος και λίγο σύντομα, για να μπορέσει να μιλήσει και ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε δύο σφαιρικές εκθέσεις. Αυτή την έκθεση και προηγούμενα του συναδέλφου, από πλευρά συναδέλφου Σάντρα. Δεν θα ήταν τώρα η χρονική στιγμή, ή τρεις έχουμε, εντάξει, έστω. Δεν θα ήταν τώρα η χρονική στιγμή να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για το νομικό πλαίσιο που αρκετοί ανέφεραν, πως θα έπρεπε να διαμορφωθεί. Και για μια ενιαία εσωτερική αγορά για τους πολίτες μας και δεν έχω μόνο υπόψη κάποιες επιμέρους διατάξεις που είναι προς όφελος των πολιτών μας και επιμέρους θέματα για την κοινωνική συζήτηση, αλλά έχω υπόψη περισσότερο μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι οι πολίτες μας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποια είναι αυτή η ενιαία εσωτερική αγορά για αυτούς και τι δίνει ως κέρδος. Γνωρίζουν μόνο επιμέρους εκδηλώσεις, επιμέρους θέματα, επιμέρους ρυθμίσεις, τι κάνουμε εμείς δηλαδή για αυτά τα θέματα, για αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά, ως μία κοινοβουλευτική επιτροπή από 20 άλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τι γίνεται με την νομική επιτροπή, παρότι συνδυαζόμαστε πολύ στο έργο μας μαζί τους, ούτε ξέρουν τι γίνεται από την Επιτροπή Μεταφορών. Πώς θα δώσουμε στους πολίτες ε, μία γνώμη και άποψη και στοιχεία πώς λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Πολύ απλή ερώτηση. Από το 1957 έχουμε το στόχο Τη κοινή ενιαία εσωτερική αγορά που διατυπώσαμε στη συνθήκη για, την Ευρωπαϊκή, για τις ευρωπαϊκές οικονομικές κοινότητες. Και τότε είχαμε δασμούς, τελωνιακούς δασμούς και τα λοιπά μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης και ένα μετά το άλλο άρχισαν να καταργούνται και ένα μετά το άλλο άρχισε να δίνει μια ανάπτυξη. Έχουμε μια εξαιρετική διατύπωση που μετά και από 20 και παραπάνω χρόνια πώς περάσαμε από την κοινή αγορά στην ενιαία εσωτερική αγορά. Οι ελευθερίες που δίνονται στους πολίτες και που θέλουμε να διασφαλιστούν. Ελευθερία κυκλοφορίας των ατόμων, των αγαθών, της παροχής υπηρεσιών και ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Και όλα αυτά είναι αυτονόητο. Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε κάτι πρέπει να είναι φιλικό Κά, όλα αυτά προς την κοινωνία και στους πολίτες. Δεν κάνουμε νομοθετήματα για κράτη, ούτε για το Ευρωκοινοβούλιο. Κάνουμε νομοθετήματα και νόμους για την ενιαία εσωτερική αγορά για τους πολίτες, ώστε να απολάβουν αυτών των ελευθεριών οι πολίτες με τον καλύτερο τρόπο και όλα τα οποία δεν είναι φιλικά προς τους πολίτες και φιλικά προς την κοινωνία θα ήταν λανθασμένα και δεν θα ανταποκρινόντουσαν σε αυτή την εντολή. Και τώρα όταν έτσι σφαιρικές εκθέσεις επί συνολικών θεμάτων έχουμε και προβληματιζόμαστε επ' αυτών, δεν θα ήταν η χρονική στιγμή και συγκυρία να προβαίναμε σε μια ιεράρχηση και ένα τη δόμηση ενός νομικού πλαισίου που θα είναι κατανοητό και για μας και για τους πολίτες. Γιατί είμαι πεισμένος ότι αν μας ρωτήσει κάποιος εξηγήστε μου κύριε την ενιαία εσωτερική αγορά τότε θα εξηγήσουμε τα δικά μας θέματα που μας απασχολούν αλλά όχι την ενιαία εσωτερική αγορά και σε όλους συμβαίνει αυτό. Και ρωτώ με, διαρωτώ με, είναι αυτό πραγματικά το σωστό και σημαντικό στο τέλος τέλος να μην μπορούμε να διαρθρώνουμε τα πράγματα έτσι ώστε τα μεγαλύτερα θέματα όπως η απελευθέρωση, οι, διάφορες ελευθερίες που θέλουμε να διασφαλιστούν για τους πολίτες να μην μπορούν να επεξηγηθούν. Πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα να επεξηγήσουμε αυτά τα θέματα μέσα σε ένα πλαίσιο ε, ουσιώδες που θα προβαίνει σε αυτή τη ρύθμιση όταν λέμε ελευθερία του ατόμου, των ατόμων, σε αυτό φυσικά ανήκουν και τα θέματα της υγείας. Όταν μπορεί να κυκλοφορεί κανείς ελεύθερα μέσα σε μια αγορά, πρέπει και για την υγεία του να μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Όταν κάνουμε λόγο για την ελευθερία κυκλοφορία των αγαθών, φυσικά εννοούμε και την ε, δυνατότητα ενός συνετού λογικού πλαισίου για την ε, αγορά προϊόντων, προστασία καταναλωτών. Όταν κάνουμε λόγο για την περιπαροχή υπηρεσιών τη ελευθερίες, για τις ελευθερίες πρέπει να δούμε τι γίνεται και στις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να μπορούν οι πολίτες να εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία. Έχουμε λοιπόν την οδηγία περιπαροχής υπηρεσιών αλλά έχουμε και την ελευθερία για τα θέματα μεταφορών. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για αυτά, αλλά πρέπει οι πολίτε να γνωρίζουν τι γίνεται και για τι μεταφορέ. Το ίδιο ισχύει και για τι ελευθερίε κυκλοφορίε των κεφαλαίων. Είμαστε αρμόδιοι για θέματα προστασία των καταναλωτών και ε, εν μέρη ε, συναρμόδιοι για θέματα ε, πιστώσεων και δανείων προ του καταναλωτέ. Αλλά αυτά ρυθμίζονται στα θέματα τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Πρέπει να ξέρουν οι πολίτε τι γίνεται σε σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, Πιστεύω ότι θα έπρεπε να προβληματιστούμε για όλα αυτά τα θέματα όταν έχουμε τέτοιε εκθέσει. Αν θα μπορούσαμε να τα καταφέρναμε για την ενιαία εσωτερική αγορά που δεν καλύπτεται μόνο από τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή αλλά είναι συναρμόδιε όλε οι άλλε Κοινοβουλευτικέ Επιτροπέ του Κοινοβουλίου να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα προ του πολίτε. Συνεμπλέκονται και άλλε Κοινοβουλευτικέ Επιτροπέ και πρέπει να ε, υπάρχει ένα σφαιρικό πλαίσιο. Χωρί να επισέθω σε λεπτομέρειε θα ήθελα μόνο ένα μικρό παράδειγμα να δώσω και να τοποθετηθώ εγώ έτσι υπέρ τη ενιαία εσωτερική αγορά ως ενό νομικού πλαισίου, μιας νομικής τάξη πραγμάτων που θα μας βοηθήσει να πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα ιδέα και από ό,τι βλέπω είστε ε, έχετε κάθε δικαίωμα να υποβάλλετε μια σχετική πρόταση. Φιλόδοξη ίσως να είναι πιο κοντά στην έκθεση της κυρίας Καρνιέτε, να ταιριάζει περισσότερο στο, στην έκθεση Καρνιέτε. Θα ζητήσω τώρα από την εκπρόσωπο της Επιτροπής να κάνει κάποια σχόλια και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Κορέιντε Κάμπος και μετά θα περάσουμε στην έκθεση που ζωή. Έχουμε ακόμα μία ώρα. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τη συζήτηση και τις προτάσεις για τη τμήμα αυτό της, ε, του νομοθετικού κειμένου για την ενιαία αγορά. Πολύ σημαντικό όπως αναφέρατε και εσείς για την Επιτροπή. Εμείς ζητούμε επαναπροσανατολισμό των πολιτικών της ενιαίας αγοράς και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις πληροφορίες και στο feedback που παίρνουμε για το τμήμα αυτό να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που τέθηκαν από την κυρία για παράδειγμα για την, τον έλεγχο της υπεύθυνη ενημέρωσης, ε, της υπεύθυνη, του υπεύθυνου δανεισμού. Εμείς έχουμε στόχο την προστασία του καταναλωτή, άρα η έμφαση στη δράση αυτή δεν θα είναι αυτή που προτείνει το κείμενο της δράσης αυτή τη στιγμή, αλλά θα δίνει μεγαλύτερη, θα εστιάζεται περισσότερο στην πρόληψη των προβλημάτων των δανειοληπτών, αλλά γενικότερα των προβλημάτων στον τομέα αυτό το χρηματο, της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ακριβώς για την πρόληψη κρίσεων όπως αυτών που ανέκυψαν στις ΗΠΑ, για παράδειγμα εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή της ε, πρότασης. Φέτος θα υποβληθεί από την Επιτροπή ένα μεγάλο σημαντικό κείμενο που το θεωρούμε παράλληλα με την πρόταση για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίε. Ε, εξίσου σημαντικό κείμενο και αυτό για την ενδεδειγμένη προστασία των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τις ε, συμβάσεις, τις δημόσιες συμβάσεις. Εμείς προβαίνουμε σε βαθύτατη αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Θα εξετάσουμε την κατάσταση του πώς οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος ε, ανατίθενται σε τρίτους, σε ιδιώτες. Αυτό και είναι ένα θέμα που θα θέσουμε σε συζήτηση γενικότερα στο πλαίσιο των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί στο τέλος του έτους από την Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα. Ξέρω τις συζητήσεις που υπάρχουν για το αν χρειάζεται να υπάρχει ένα κείμενο πλαίσιο για τις υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ε, απλά σας λέω ότι υπάρχει κινητικότητα δεν είμαστε ε, ακινητοποιημένοι. Απλά περιμένουμε να δούμε πώς θα αξιολογηθεί η δράση αυτή και αν χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο. Για τον κοινωνικό αντίκτυπο, μια πολύ δύσκολη βέβαια θέση, η κοινωνική ρήτρα ιδίω. Θέλω να υπογραμμίσω ότι στην Επιτροπή αγωνιζόμαστε για να κάνουμε ένα μια σωστή αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η αξιολόγηση στο εσωτερικό της υπηρεσίας συνεχίζεται προσεκτικά. Έχουμε εξετάσει ε, τις λεπτομέρειες. Είναι δύσκολη δουλειά και τον, ε, στην αξιολόγηση αντικτύπου θα εξετάσουμε βέβαια και τον αντίκτυπο στη, στην απασχόληση. Καταλαβαίνω τις συζητήσεις που διεξάγονται, τις ε, καλωσορίζουμε γιατί εμείς τις ξεκινήσαμε μεταξύ άλλων, αλλά λάβετε υπόψη ότι θα υπάρξει βελτίωση στο μέλλον και στην Επιτροπή θέλουμε να διεξάγουμε σωστούς ε, ελέγχους κοινωνικού αντικτύπου. Αυτά προς το παρόν. Στην πρόταση 41 λέτε πως η Κομισιόν μέχρι το Φεβρουάριο του 2011 θα υποβάλει μία, οδηγίους, μία οδηγία για ενιαία αγορά στεγαστικών δανείων. Για μένα μοιάζει κάτι το διαφορετικό εδώ πέρα. Πως θέλετε την απελευθέρωση αυτής της αγοράς, κάτι το οποίο βέβαια είναι διαφορετικό από οδηγία προστασίας των καταναλωτών και ναι, ε, έχετε πει όμως πως θα είναι πολύ αργότερα από το Φεβρουάριο 2011. Όπως προσπάθησα να πω, όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά, δεν θα είναι αυτή η έμφαση που θα δοθεί στην νομοθεσία, θα έχουμε, δώσουμε περισσότερο βάρος στην προστασία των καταναλωτών. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον εισηγητή για να κάνει ίσως κάποιες ε, τελευταίες παρατηρήσεις, Αντώνιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους ε, για τον πλούτο των παρεμβάσεων που έκαναν και τον πλούτο επίσης ε, και την ζωντάνια των επικρίσεων που έκαναν. Αισθάνομαι κάπως όπως ο Επίτροπος Μπαρνιέ όταν για παράδειγμα κατηγορούμε εμείς ε, το έγγραφό του, την ανακοίνωσή του των σημείων αυτών ότι είναι απλώς ένα εμβαλωματικό συνονθήλευμα και μας απαντά ότι είναι το καλύτερο που ήταν δυνατόν να επιτευχθεί στο, στη συνεργασία 12 ή 13 επιτρόπων και γι' αυτό αυτή η κατάρα στην αποκαλέσω έτσι να συντάσσουμε μια έκθεση ή να αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα το οποίο διεισδύει και ε, ε υπησέρχεται σε τόσες διαφορετικές ε, πλευρές και παιδεία και σε τόσα, τόσες διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο είναι μια κατάρα που μας ε, διώκει και μας καταδιώκει κατά την επιτέλεση του έργου μας. Θα υπάρχουν πάντα επικρίσεις όσον αφορά την προσέγγιση που υιοθετούμε ή ότι είναι πολύ γενικόλογοι ή ότι θα πρέπει να εξεταστούν 50 θέματα σημείο προς σημείο ή ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί συνέχιση διότι είναι κατακαιρματισμένη η προσέγγιση κτλ. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, να συμβιώνουμε με αυτή την ε, ας το πω έτσι πολυμορφία ζητημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τόν προσωπικά και εκ νέου να ευχαριστήσω για τις επικρίσεις που κάνει, για την δομή που έχω υιοθετήσει, τη διάρθρωση για τη βάση αυτών των επικρίσεων και που, γιατί το ότι είχαμε εγκρίνει μια τριπλή προσέγγιση που θα υιοθετείται από όλες τις τρεις εκθέσεις και για το τι συμβαίνει με τη δική μου έκθεση θα συγχωνεύσουμε αυτό το θέμα όσον αφορά τα κένα, όσον αφορά τα common principles and values θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο που θα αποκαλούμε γενική αξιολόγηση, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, θέτοντας τους Ευρωπαίους πολίτες στην καρδιά της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, που είναι αν θέλετε, μετατροπή ε, κυριολεκτικά της πρότασης της Επιτροπής και ε, ε, εφαρμογή εδώ. Θα έχουμε λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες που θα πρέπει να εξεταστούν και βραχυπρόθεσμα. 100% συμφωνούμε με τη συνάδελφο και πρέπει μόνο να ευχαριστήσω για αυτά που είπε, για τις προτάσεις που διατύπωσε. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι ολοκληρώνονται εδώ οι συμφωνίες μας σε αυτά τα θέματα. Αφενός για λόγους ε, ανεπαρκούς πληροφόρησης. Από την άλλη πλευρά λόγω διαφορών ιδεολογικών και διαφορών απόψεων οι διαφωνίες είναι μεγάλες ε, οι διαφορές. Από πλευράς της κυρίας Τόιν μου ασκούνται επικρίσεις επειδή λέει δεν υπάρχει μια σαφής ε, ταύτιση και εντοπισμός ιεραρχήσεων προτεραιοτήτων μα είναι πέντε οι προτεραιότητες αυτές βραχυπρόθεσμα short term για τη στρατηγική μας. Αυτές είναι οι πέντε προτεραιότητες με τη σειρά ιεράρχησης, με τη σειρά που απαριθμούνται και παρουσιάζονται. Ίσως εδώ θα μπορούσα να δεχθώ ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι πιο γενικόλογοι, πιο σφαιρικοί και πιο είναι ευρύτεροι. Όλες οι άλλες όμως είναι απορρέουν από επιμέρους σημεία e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο, καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης και πειρατείας, μια πολιτική επικοινωνίας που θα είναι αποτελεσματική και ένα σύστημα αξιολόγησης σύστημα αξιολόγησης όσον αφορά την υλοποίηση των κοινωνικών θεμάτων. Το να είναι πιο εξειδικευμένο κανείς ε, από αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ίσως θα είναι δυνατό να είναι πολύ δύσκολο να είναι κανεί πιο εξειδικευμένο. Επίσης όταν αναφέρει συνάδελφος Τσούιν ε, και αναφέρει ότι και λέει ότι η κοινωνική λέει ρήτρα, η οριζόντια, εγκάσια είναι δύσκολο, δύσκολο να επιτευχθεί. Μα αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία μας όμως, σε συνταγματικό πλαίσιο και βρίσκεται στη σελίδα 19 της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πρέπει εδώ να το παρανοούμε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποβάλουμε προτάσεις. Πώς είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αυτή η προσέγγιση. Και ακριβώς εδώ έχουμε τον αριθμό 5, τον, την πέμπτη πρότασή μου ως προτεραιότητα στην απαρίθμηση των προτεραιοτήτων. Ένα σύστημα benchmarks, βέλτιστων ρητρών και προδιαγραφών στις οποίες θα ανταποκρινόμαστε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που ακριβώς αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα, για το τι θα πρέπει να γίνει σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να πω στην κυρία Τόιν. Είναι δυνατό και εφικτό να γίνει αυτό και είναι προτεραιότητα. Εντάξει, είναι προφανές ότι να ακολουθήσει κανείς και είχα ένα πρώτο πειρασμό να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τις 19 προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να τις σχολιάσω κιόλα. Αλλά να ακολουθήσουμε αυτές τις 19 προτάσεις τι θα ήταν. Θα ήταν να ευθυγραμμιστούμε σε μια ας το πω έτσι επίκριση, στις επικρίσεις που εμείς ασκούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήθελα να βασιστώ καλύτερα σε μια ολιστική, σφαιρική προσέγγιση που θα δίνει μια άλλη επικέντρωση αναγνωρίζω ότι καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά στη συγκυρία των gaps τώρα και πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά σε ένα ενιαίο κεφάλαιο και ότι τώρα έχουμε το περιορισμό του εύρους που τίθεται σε σχέση με την έκθεση όσον αφορά αριθμό σελίδων και ε, τυπογραφικών χαρακτήρων θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολλές από αυτές τις προτάσεις ε, αν όχι όλες που δεν είναι δυνατόν να τις εντάξουμε σε αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ εν πάση περιπτώσει την κυρία συνάδελφο Τόιν για τις προτάσεις της, για τις κριτικές της ακόμα και τις επικρίσεις της. Σε σχέση με τον συνάδελφο Κρόιτσμαν πρέπει να πω ότι για τις προτεραιότητες ήδη έχω απαντήσει. Για το θέμα της ενέργειας και της ψηφιακής, ε, του ψηφιακού θεματολογίου επίσης πιστεύω ότι έχουν διευθετηθεί, έχουν απαντηθεί. Ικανοποιούμε διαπιστώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία σε σχέση με τις συλλογικές δράσεις. Δεν πρέπει να συμφωνούμε απλά για να συμφωνούμε. Εδώ έχουμε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτά, έπρεπε να τοποθετηθούμε. Δεν, έπρεπε να, δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε κάποια στοιχεία και να ασχοληθούμε απλά με άλλα. Για την κυρία Ρούιλε ανέφερε πολλά κενά λέει που υπάρχουν πράγμα που φυσικά πιστεύω με τη βοήθειά της ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε με τις σωστές τροπολογίες. Είναι προφανές ότι αναφέρω τον επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλά έχοντας μελετήσει τις προτεραιότητες ε, ευρύτερα το roaming, η περιαγωγή και η ευρυζωνική προσέγγιση που ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διάδοση δεδομένων. Όσον αφορά το θέμα για τις, ε, τα ενυπόθηκα δάνεια, εδώ υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις στη συνέχεια για αυτό το θέμα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία ο τόνος, ο γενικός τόνος αυτών των παρεμβάσεων είναι ότι αφενός είναι δύσκολο να υπάρξει ένας εναρμονισμός μεταξύ όλων των χωρών όσον αφορά τα θέματα ενυπόθηκων δανείων. Από την άλλη πλευρά όμως κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αιώνια σε αυτή την κατάσταση εις το διηνεκές του να είμαστε ευάλωτοι και εύτρωτοι σε οποιαδήποτε νέα ας το πω δυσλειτουργία της αγοράς και οποιοδήποτε νέο πρόβλημα. Γι' αυτό ε, υπάρχει η, παρα... η υπονόμευση της οικονομικής ισορροπίας και το είδαμε αυτό ότι συνέβη. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το γεγονό ότι αυτό είναι θέμα συγκεκριμένη αρμοδιότητα άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών μα κάνει να σκεφτούμε στο σφαιρικό χαρακτήρα που πρέπει να υιοθετήσουμε στην προσέγγιση μα. Συμφωνώ ότι εδώ απουσιάζει μια αναφορά στι κλιματικέ ε, αλλαγέ και στην κλιματική κρίση. Όπω επίση και για τα ε, κοινωνικά θέματα πρέπει να αναφέρουμε και τι κλιματικέ αλλαγέ. Ε, από τον Μάκομ Χάρμπορ και τα σχόλιά του τώρα. Ήδη ανέφερα έδωσα μια απάντηση για τα δάνεια, ε, για τις υπηρεσίες συνολικού ε, καθολικού συμφέροντος ε, που πρέπει να ενταχθούν ε, σε σχέση με τα σχόλια που έγιναν μέσα στην απάντηση που θα δώσουμε το ότι επί τόσα χρόνια κινούμαστε προς τα εδώ και προς τα εκεί αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθεί μια πολιτική απόφαση για την οδηγία πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο είναι ουσιώδου σημασίας και αληθεύει αυτό πράγματι εγώ πιστεύω ότι φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση είναι όμως πολύ σημαντική κάθε χώρα διατηρεί τις παραδόσεις στην ιστορία της, στο παρελθόν της, όλα αυτά καμιά φορά υπάρχουν, υπάρχει και το ελεγκτικό συνέδριο ή το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που αποφασίζει και τολμά να λάβει αποφάσεις που δεν είναι ευχάριστες ούτε για τους μεν ούτε για τους δε. Αναγνωρίζω λοιπόν, είναι αναγκαίο, είναι θεμελιώδες να αποφασιστεί αυτό το, να ρυθμιστεί αυτό το πλαίσιο, αυτό το θέμα. Και όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά για τους πολίτες, συμφωνώ απόλυτα με τον Μάκομ όταν λέει για τις πληροφορίες και ότι πρέπει να υπάρχει εδώ στον πίνακα των προτεραιοτήτων να ενταχθεί η ανάπτυξη σωστής πολιτικής επικοινωνίας σε σχέση με την ενιαία εσωτερική αγορά που θα λαμβάνει υπόψη τα, τα, θέματα πολιτικής που έχουν επίπτωση στη ζωή των πολιτών. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την επικοινωνία για ενημέρωση των πολιτών. Τέλος, υπάρχει ένα σημείο που έχει δίκιο ο Μάκομ Χάμπος στις επικρίσεις που ασκεί λέει ότι η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει πιο επίμονα τον στόχο της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είναι μια απόλυτα αντικειμενική κριτική αυτή η επίκριση που την δέχομαι 100%. Είναι προφανές ότι αναφέρω το ζήτημα της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μην χάσουμε θέσεις απασχόλησης. Αυτό όμως είναι αμυντικού χαρακτήρα. Συμφωνώ όμως με το Μάκομ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην έκθεση ε, και με τροπολογίε μπορεί να γίνει αυτό, να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην δημιουργία θέσεων απασχόληση στην έκθεσή μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Συμφωνώ. Σε σχέση με τα σχόλια που έγιναν από την Evelyn Γκέπχαρτ, την Barbara Βάιλερ Νομίζω ότι ήδη αναφέραμε τα θέματα που αναφέρονται σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα, την παροχή υπηρεσιών, τα επαγγελματικά δικαιώματα και κατάρτιση με, τα, με την κατοχήρησή τους που πρέπει να ενταχθούν και αυτά. Εν τέλει θα ήθελα να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω για την παρέμβαση του συνα, συναδέλφου Μάιερ. Και αυτό γιατί λέει ακριβώς αυτό το οποίο εμείς ε, πρέπει να δώσουμε μάχη και θέλουμε να δώσουμε μάχη. Δύο πράγματα. Πρώτον, νομικό πλαίσιο. Να ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο. Να μην φοβόμαστε να το δημιουργήσουμε και να το προαγάγουμε. Δεύτερον, συζήτηση για τα κοινωνικά θέματα. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Η κοινωνική, ο κοινωνικός προβληματισμός νομιμοποιείται και είναι θεμητός. Και να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την έννοια της ελευθερίας στην ενιαία εσωτερική αγορά. Πρέπει ακριβώς προς και εξυπηρέτηση των πολιτών που μας εκλέγουν και είμαστε εκπρόσωποι τους εδώ να ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα και ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια που θα μπορέσετε να μας δώσετε με τροπολογίες από πλευρά σας. Και ήδη αναφέρθηκα εν παρόδο στα σχόλια της Επιτροπής για τα δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια και για τις ε, οικονομικές υπηρεσίες γενικού καθολικού συμφέροντος. Ευχαριστώ, ολοκλήρωσα. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Uh, well, now going to... Ευχαριστώ για τα σχόλια σου. Τελευταία έκθεση του Κρίστιαν Μπουζόη. Θα ήθελα ε, ένα ε, ημίωρο συζήτηση και δέκα λεπτά για την σύνοψη. Θα έρθει ο κύριος Κάρας, η κυρία Ρούλα είναι εδώ καλύπτα πάντα, η υπάρχει... Υπάρχουν οι άλλοι σκιώδεις. Υπάρχει κάποιος άλλος σκιώδης που θέλει να μιλήσει για την έκθεση αυτή. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κλείνω τον κατάλογο. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο από τα καταληκτικά συμπεράσματα και κατόπιν θα μιλήσει και η Επιτροπή. Συνάδελφοι, να είστε κάπως ε, συνοπτικοί. Η κυρία Βανιό αν θέλει να ξεκινήσει τη συζήτηση από τους Κιώδης. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσόη, διότι πραγματικά συνεργαστήκαμε πολύ στενά σε πολλές συναντήσεις ε, που κάναμε. Αυτό που θεωρώ σημαντικό για την έκθεση είναι κάποιες προτεραιότητες εξίσου σημαντικές και για τις τρεις εκθέσεις. Κύριε Μπουζόη, στην έκθεση για την οποία σας συγχαίρω έχετε μια σαφή δομή με ξεκάθαρες θεματικές, ξεκάθαρες προτεραιότητες, έστω και αν, τέλος πάντων το ξανασυζητήσουμε, εγώ δεν θα είχα ακολουθήσει την ίδια δομή. Διότι πιστεύω ότι το τμήμα 3 και το τμήμα 4, αγορά για τις επιχειρήσεις και αγορά για τις υπηρεσίες, περιλαμβάνουν δομές, υπηρεσίες, αλλά περιλαμβάνουν και πολίτες και επιχειρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δύο αυτά κομμάτια είναι τα πιο σημαντικά στην έκθεσή σας. Προφανώς καινοτόμως είναι η αγορά, προφανώς η ψηφιακή αγορά. Επανέρχομαι στη δομή σας πάντως. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και οι τροπολογίες που θα υποβάλω ως ομάδα προς τα εκεί θα τίνουν. Στο πρώτο τμήμα καινοτόμως είναι η αγορά πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ουσιαστικά τη σπουδαιότητα της ε, ενίας αγοράς, το 6 και το 7 και τα κριτήρια που θέλουμε να θέσουμε. Τα κοινωνικά δε κριτήρια είναι πολύ σημαντικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους ώστε να προστατευτούν και να προστατευτούν όταν μπαίνουν στην, ε, ε στις δημόσιες συμβάσεις που μπαίνουν συχνά ως υπεργολάβοι. Είναι σημαντικό λοιπόν επίσης να διευκρινίσουμε και τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Ζούμε σε μια χρονική στιγμή μάχης κατά τη αλλαγής του κλίματος. Είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες αγορές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σαφή κριτήρια που θα τους επιτρέψουν να λύνουν τα ζητήματα με ασφάλεια δικαίου. Κάτι επίσης που δεν αναφέρει το κεφάλαιο αυτό και θεωρώ σημαντικό. Να υπάρχει μία μνήμα στις επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και μεταφορών. Μέσω των ΣΒΙΤ, το είπε ο Μάλκομ, και έτσι μπαίνω στο δεύτερο τμήμα σας. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε. Μιλάτε για την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Τι εννοείτε να δημιουργηθεί μια, ένας, μια πραγματικά καθολική υπηρεσία. Πολύ σημαντικό. Προφανώς προτεραιότητες, το τρίτο τμήμα, δεν θα σας ε, εκπλήξει αυτό, το τραπεζικό κλάδο. Κάτι που συνδέεται και με τις προηγούμενες εκθέσεις, ιδίως του κ. Κορέιέντε Κάμπος. Και εδώ θεωρώ σημαντικό και για τις μικρές επιχειρήσεις και για τους πολίτες να διευκρινίσουμε πραγματικά τους κανόνες της τραπεζική, του τραπεζικού κλάδου και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, ούτω ώστε να υπάρξει αν όχι εναρμόνιση, τουλάχιστον κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ χωρών και στο εσωτερικό χωρών μερικές φορές, ανάλογα με τις περιφέρειες. Είναι σημαντικό λοιπόν να διευκρινίσουμε το δρόμο που θέλουμε να χαράξουμε και τα όρια που δεν πρέπει να υπερβούμε. Κατόπιν, δεν θα σας εκπλήξει πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε όταν μιλούμε για ανάπτυξη πολύ μιλούμε και σωστό είναι ανάπτυξη σημαίνει και θέση και δημιουργία θέσεων εργασία. Προφανώ μέσω καινοτομία, μέσω υπηρεσιών και εδώ Μάλκολμ οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και οι υπηρεσίες οικονομικού Όλοι Σχολιάστηκαν επί μακρόν σήμερα. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε νομικό πλαίσιο που θα δεσμεύει τα πάντα. Όχι, προφανώ. Ωστόσο, κύριε Κοράτσα Μπίλτ, ε, θα σας ε, το σχολιάσετε. Τι εννοείτε με τον όρο απορρίθμιση. Αν μπούμε σε ένα τέτοιο σύστημα, νομίζω ότι πηγαίνουμε στον αντίστροφο δρόμο από αυτό που θέλει ο πολίτης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίε λοιπόν κοινή ωφέλεια και, καθολικής και, γενικής, και γενικού οικονομικού συμφέροντο ε, καθορίζουν εκ νέου είναι σημαντικέ γιατί πρέπει να καθορίσουν τι αξίε που θα περάσουμε. Ε, μην ξεχνάτε ότι οι υπηρεσίε αυτέ βοήθησαν την απάλυνση του αντικτύπου της κρίσεως και σε κάθε περιοχή εξασφαλίζουν κοινωνική συνοχή, υπηρεσίες προς όφελον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προφανώς σε σχέση με την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές, ε, ΣΒΙΤ κλπ. Ιδίω στις διασυνοριακές ζώνες, στο δεύτερο κεφάλαιο, νομίζω εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα να προσθέσουμε. Συνολικά, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως κάτι που θεωρώ ότι λείπει στο τέταρτο τμήμα. Σε όλες τις διασυνοριακές ζώνες είναι σημαντικό να φροντίζουμε να υπάρχει η καλύτερη και πιο προσαρμοσμένη δυνατή υλοποίηση της οδηγίας υπηρεσιών σε συνδυασμό, το είπε και ο Πρόεδρος, με την επερχόμενη ε, οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Είναι σημαντικό το να φέρει ο κύριος Μπουζόη στο σημείο 20 είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Χθε ήμουν σε μια συνάντηση στην Επιτροπή με τον κύριο Τίτζε που είναι ο υπεύθυνο του θέματος, όπου συζητήσαμε με επαγγελματίες, φαίνεται ότι είναι πιθανό σε κάποια επαγγέλματα να υπάρξει ένα, μια ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα που θα εξασφαλίζει και τον ε, καταναλωτή και τον, ε, τον ελεύθερο επαγγελματία που θα συνάδει με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Και στο σημείο αυτό χρειάζεται μια μεγαλύτερη διευκρίνηση, τουλάχιστον μέσω τροπολογιών. Πάντως εδώ πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα καλό πακέτο και με τις προτεραιότητες ε, που τίθενται και στις άλλες δύο ε, εκθέσεις. Και πρέπει να σας πω κύριε Κανίατε ότι πραγματικά εκτίμησε ιδιαίτερα τις, ε, την έκθεση με δύο-τρεις αλλαγές. Τώρα η συζήτηση, οδηγία, κανονισμός, εντάξει να τα συζητήσουμε. Ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κανονισμούς μόνο και μόνο για να έχουμε κανονισμούς. Οι πολίτες λένε συχνά όχι πολύ νομοθεσία. Ε, λιγότερη νομοθεσία, μεγαλύτερη ποιότητα. εντοπίζοντας σωστά τις προτεραιότητες και τις ανάγκες όλων των επιπέδων. Με αυτέ τι ε, κατευθυντήριε γραμμέ που παρουσιάζουμε στα τελειοδοσία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε με την Επιτροπή και ελπίζω το Συμβούλιο να συμφωνήσει στι γενικέ γραμμέ, γιατί πρόκειται για καθοριστική σημασία κείμενο άλλωστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά τα οποία κάνετε για την αμοιβή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που θα είναι επίσης πολύ σημαντικό κατόπιν. Ο Ότμαρ Κάρα έχει έρθει. Αν θέλει τον λόγο θα τον παρακαλέσω να μιλήσει ω και ο του ΕΛΚ στην έκθεση Κύριε Πρόεδρε, κύριε κυρίε και κύριοι, συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων έχουμε την ε, ακρόαση με τους νέους επικεφαλείς ε, τραπεζών και εποπτικών αρχών και ασφαλιστικών εταιριών. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να συγχάρω τον συγητή. Έχω όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις οποίες θα καταθέσουμε και τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα στο άρθρο 9 μιλάμε για τη σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο που αναφέρεται ως ε, εμπόδιο στην εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων. Το απόγευμα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, θα ψηφίσουμε για την οδηγία δικαιωμάτων των καταναλτών και θεωρώ πως θα πρέπει να περιμένουμε και να αξιολογήσουμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το φιλόδοξο έργο πριν περάσουμε στο επόμενο βήμα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δούμε πως θα υπάρχει ενιαίο δίκαιο των συμβάσεων εάν υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, άρθρο 13 όπου μιλάμε για τις πληροφορίες. Νομίζω πως θα πρέπει το βάρος να πάει σε όσο δυνατόν πιο συνοπτικές ε, πληροφορίες που θα δίνονται από, ένα, από μια υπηρεσία, από ένα γκισέ. Δεν είναι το θέμα μόνο η επέκταση, αλλά και η σύνοψη, η διαφάνεια, η σαφήνεια και το ποιος δίνει τις πληροφορίες. Τρίτον, για την διαδικασία δημοσίων προμηθειών. Εδώ πέρα απαιτείται βεβαίως αποτελεσματικότητα και ευελιξία, αλλά στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη θέση των υπηρεσιών των κοινοφελών. Τέταρτον, άρθρο 18 που αφορά θέμητες εμπορικές ε, πρακτικές. Εδώ πέρα πάρα πολλοί θεωρούν πως έχει συνταχθεί πάρα πολύ στενά γιατί δεν είναι μόνο οι μικρόμεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 2008 είχε ζητήσει από την Κομισιόν να κάνει κάτι για την παραπλανητική διαφήμιση δυστυχώς, από εταιρείε που στέλνουν στους πάντες Δυστυχώς ε, δεν έχει γίνει τίποτα και εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Πέμπτο, στον τομέα των ε, αντιπροσωπιών υπηρεσιών, από πω πως το Κοινοβούλιο το 2009 διακομματικά αποφάσισε κατά μιας πανευρωπαϊκής ρύθμισης. Εμείς θεωρούμε πως το τωρινό νομικό πλαίσιο είναι επαρκές. Ισχύουν οι γενικές αρχές ε, της ε, Σύμβασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης, διαφάνεια, ίση μεταχείριση, η απαραίτητη ευελιξία και ο αγώνας και βεβαίως καταπολέμηση της τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Επίσης, δεν έχουν οριστεί ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα χρειαζόταν να κάνουμε. Επίσης θα ήθελα να σκεφτείτε πριν ε, καταλήξουμε σε ένα νέο έντυπο, νέα ταυτότητα περί επαγγελματικών προσώπων να αξιολογήσουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία ενός προστιθέμενου εγγράφου αυτή τη στιγμή. Επιπλέον πρέπει να πάμε σε μια ενίσχυση των επιχειρήσεων η οποία θα γίνει μέσω σύνδεσης των ε, επιχειρηματικών μητρών. Είναι καλή λοιπόν η έκθεση και είμαι πεπισμένος πως με αυτή την έκθεση θα μπορέσουμε να δώσουμε μια δυνατή θέση τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και να συνεισφέρουμε στην Κομισιόν έτσι ώστε η νομοθεσία περιστορικής αγοράς να αρχίσει να κινείται και να προσφέρει μια νέα δυναμική. Παρακαλώ όμως την Κομισιόν να βοηθήσει για να γίνει αισθητή αυτή η δυναμική και να μην ε, κατατμηθεί μεταξύ διαφόρων επιτρόπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ότμαρ. Κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Καλωσορίζω την ξεκάθαρη δομή και τις προτεραιότητες. Έχω και εγώ πολλές παρατηρήσεις. Ο Μάλκομ ανέφερε την δημιουργία θέσεων εργασίας στην προηγούμενη έκθεση. Νομίζω πως σε αυτή την έκθεση ταιριάζει, αναφέρθηκε και από την Κομισιόν και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά στις πολλές δυνατότητες της παράσινης τεχνολογίας, προστασίας του περιβάλλοντος, ε, να δημιουργηθούν εκεί πέρα θέσεις εργασίας και η Κομισιόν για τη νέα ανακοίνωσή της για τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχή είπε πως θα πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε λοιπόν και θα καταθέσουμε μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Κατόπιν στο σημείο 3 αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αλλά δεν αναφέρεται αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν στο τομέα της τυποποίησης και πρέπει να συμπληρωθεί είναι μια προτεραιότητα της Επιτροπής μας οπότε θεωρώ πως πρέπει να πούμε και κάτι. Κατόπιν να αναφέρω πως η Κομισιόν επίσης αναφέρει στα σημεία 8 και 10 το ζήτημα επανακαθορισμού της φορολογίας ενέργειας, οικολογικό αποτύπωμα, όλα αυτά δεν αναφέρονται αρκετά, θέλω συμπληρώσεις. Επόμενο σημείο το ανέφεραν οι προλαλήσαντες, τα πάρα πολλά μέτρα της Κομισιόν όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, εκεί πέρα θα θέλαμε μια πιο σαφή διάρθρωση. Ενδιαφέρον είναι πως από τη μία γίνεται μια αξιολόγηση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δύο νέα νομοθετικά μέτρα τα οποία προτείνονται και πώς κολλάει αυτό με την καλύτερη, ε, καλύτερη ρύθμιση όταν δεν έχει γίνει αξιολόγηση. Πρέπει να γίνει η αξιολόγηση πριν προετοιμάσουμε νέα νομοθετικά μέτρα. Αλλιώς θα υπάρξει κατακαιρματισμός στο δίκαιο των δημοσίων προμηθειών και κατόπιν προτείνει πράγματι η Κομισιόν ε, κάποια πράγματα για τις ε, αντιπροσωπείς υπηρεσιών. Δεν ξέρω. Και εδώ πέρα είπε το στο ο κύριος Καράς ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε πράγματα πριν την αξιολόγηση. Και τέλος η πρόταση 24, την οποία συζητήσαμε μόνο παρενθετικά. Εδώ πέρα προτείνει η Κομισιόν για το έτος 2011 κοινοτικό μέσο για να είμαστε σε καλύτερη θέση να έχουμε καλύτερη συμμετρία στην πρόσβαση μεταξύ βιομηχανικών χωρών και μεγάλων ε, οικονομιών. Δηλαδή το θέμα της αμοιβαιότητας και μήπως θα πρέπει να καταθέσουμε, δεν ξέρω, μια προφορική ερώτηση, ίσως στην επόμενη ολομέλεια για να ξεκαθαρίσει αυτός ο κατάλογος μέτρων της Κομισιόν. Γιατί αν γίνουν όλα αυτά μεμονωμένα θα οδηγηθούμε σε μια πάρα πολύ ασαφή δομή στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Οπότε σας παρακαλώ να ξεκαθαρίσει αυτό. Αυτά. Uh, um, Ευχαριστώ. Οι τέσσερις ομιλητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να εκφράσω τα συγχαρητηριά μου στον κύριο Μπουσό για τη δουλειά του. Όταν ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό για πρώτη φορά, βλέπουμε, από τότε που συζητήσαμε το θέμα για πρώτη φορά, βλέπουμε τεράστια ε, εξέλιξη. Κάποια γενικά σχόλια πρώτα και μετά τα ειδικότερα. Σήμερα το πρωί άκουσα όλους τους συγητές, όλες τις συζητήσεις. Είναι γεγονός ότι το θέμα της εσωτερικής, είναι θέμα της εσωτερικής αγοράς, αλλά σημαντικό. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση Μόντι, πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική. Ωστόσο κατόπιν διαπιστώνουμε ότι δεν είναι εύκολο να υλοποιήσουμε αυτά που θέλουμε ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύω, πιστεύω ότι στην Επιτροπή μας θα συμφωνήσουμε όλοι όταν όμως προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους συμπατριώτες μας τα πλονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα, ότι ανακύπτουν τοπικά ή περιφερειακά προβλήματα με τις αντίστοιχες αρχές. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε την ενιαία αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το Συμβούλιο. Να ζητήσουμε λοιπόν πολύ περισσότερο από εμά. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Ουγγρική Προεδρία να κάνει ε, δική της την εσωτερική αγορά και να την προωθήσει περισσότερο ακόμα. Ας μπω τώρα στην έκθεση Μπουσόη. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι στην τσεχική μετάφραση, αλλά Υπάρχει πρόταση εναρμόνισης των συστημάτων ΦΠΑ. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Θα δημιουργηθούν μια σειρά προβλημάτων. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπουσόη. Εδώ εμφανίζεται σαφέστερη ανάγκη μείωση τη γραφειοκρατία για τι επιχειρήσει. Αλλά στο ξεκίνημα ε, αναφέρεται αυτό. Λέει ότι επιβάλλουμε στου επιχειρηματίε μεγάλη ε, μεγάλο δημοσιονομικό βάρος, αλλά μετά αυτό δεν εμφανίζεται κατόπιν. Μία γενική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, με ενοχλεί πολύ αυτή η ιδεολογική προσέγγιση του να λέμε από τη μια μεριά τι είναι καλό για τον Ευρωπαίο πολίτη και για τους καταναλωτές και από την άλλη τι είναι καλό για τις επιχειρήσεις. Αυτή η διτή προσέγγιση είναι λάθος. Για μεθοδολογικούς στόχους όντως πρέπει να μειώσουμε τη δουλειά, να, περι, να διαιρέσουμε τη δουλειά σε τρία τμήματα, αλλά νομίζω ότι το όραμα πρέπει να είναι σαφές. Ό,τι είναι καλό για τις επιχειρήσεις δεν είναι κακό για τον κόσμο. Ό,τι είναι καλό για τον κόσμο δεν είναι κακό για τις επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Πώς ε, κάνουμε την κοινωνική Ευρώπη, πώς εφαρμόζουμε τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών όταν οι κυβερνήσει επιβαρύνονται από τα βάρη αυτά που γνωρίζουμε. Ποιος θα δημιουργήσει την κοινωνική Ευρώπη αν δεν αφαιρέσουμε από τις επιχειρήσεις τους περιορισμούς για να επενδύσουν και να προσλάβουν. Πού βρίσκεις τους πόρους για να μειώσει την ανεργία στην Ευρώπη αν δεν δώσεις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βγουν, να, να, αφαιρέσουν τις αλυσίδες που τραβάνε ακόμα. Θα ήθελα κάποιος να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Και αυτή είναι η απάντησή μου σε εσά για τον κανονισμό. Λέτε δεν θέλει ο κόσμος ρυθμιστική προσέγγιση. Αλλά από την άλλη λέτε, οι, οι, οι πολίτες μας κατηγορούν ότι υπάρχει πολύ νομοθετική ε, προσέγγιση. Αυτό είναι το πρόβλημα, όντως. Χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες και λιγότερη νομοθεσία. Λιγότερες διαδικασίες που έχουν διοικητικό κόστος και μόνο για τις επιχειρήσεις που επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Υπάρχει το Small Business Act. Ας το υλοποιήσουμε. Για την έκθεση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σκληρότερη όταν αναφέρει ότι πρέπει να φύγουν τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών που είναι η αλφαβήτα της εσωτερικής αγοράς. Το πρόβλημα, το πρόβλημα της πρόσβασης στην αγορά, στην αγορά το δικαίωμα, στο δικαίωμα εγκατάστασης. Καλό θα ήταν να, να, να υπάρξει μνήα στην ανάγκη επιβολή, όχι μόνο τι οδηγίε για τις υπηρεσίες αλλά και τι οδηγίε για τα αγαθά. Θα πρέπει να υπάρχει ε, σαφές, σαφής έκκληση για ανταγωνιστικότητα. Η λέξη ανταγωνιστικότητα εμφανίζεται μόνο ε, στην έκθεση της Επιτροπής, εκεί που λέει ότι η έκθεση ε, λέει για μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κοινωνική εσωτερική αγορά. Εκεί μόνο υπάρχει η λέξη ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να έχουμε μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Καλό είναι το small is beautiful, αλλά πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Πρέπει να ανταγωνιστούμε την Κίνα, την Ινδία. Δεν το κάνουμε μόνο με την κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ισχυρών επιχειρήσεων. Με κοινωνική ευθύνη, βεβαίως. Δεν μπορούμε ωστόσο να αγνοήσουμε τον όρο ανταγωνισμό. Και έχω δύο παρατηρήσεις που θέλω να διευκρινίσετε λίγο περισσότερο. Άρθρο 15 που λέει κοινή ε, ε, συγκρισιμότητα φορολογικών συντελεστών και κοινές κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιριών. Οι φόροι μπορεί να έχουν όντως ε, διακριτική, να, αποτελούν σημείο διάκρισης για την εγκατάσταση των ε, επιχειρήσεων και άλλες νομοθεσίες μπορεί να έχουν διακριτική διάσταση. Το σημείο 18. Τώρα, το σημείο 18 θα ήθελα να ξέρω τι εννοείται με τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα για να προστατευθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα που βάζουμε ε, στην έκθεση άμα δεν το ε, ε, εξετάσουμε προσεκτικά. Αυτά κύριε, κύριε Πρόεδρε ομαδική, ομαδικά λειτουργεί η Προεδρία. Ο κύριος Κορέιντε Κάμπος θέλει μια... Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Μια και η συνάδελφο Κοράτσα Μπίρτ άμεσα αναφέρθηκε στην έκθεση, νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσω και να πω δύο λόγια. Τρία παραδείγματα ανέφερε. Μικρότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση, περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση, ευφιέστερος εναρμονισμός και η ε, δράση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Ευθυγραμμίζομαι 100% με τις προτάσεις της. Τώρα, εκείνο το οποίο οι Ευρωπαίοι δεν χρειάζονται και δεν χρειαζόμαστε είναι απορρίθμιση, η οποία δεν θα είναι ευφυής. Δεν είναι ευφυής. Η απορρίθμιση που δεν είναι ευφυής είναι περιττή, περιτεύει και κανείς κανείς στις τελευταίες συζητήσεις δεν ανέφερε ή δεν σκέφτηκε και είπε ότι αυτό που είναι καλό για τις επιχειρήσεις ή τις εταιρείες, είναι φυσιολογικά και κατά κανόνα κακό για τους πολίτες. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο, εντάξει. Λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα. Πιθανώς ε, κακή ερμηνεία αυτών που έχουν ε, διατυπωθεί γραπτός είναι αυτή. Και ε, δεν με γνωρίζετε καλά κυρία Κοράσα Μπίρτ, αλλά θα ήθελα να σας πω και να γνωρίζετε ότι εδώ εγώ. Ήμουν ο υπουργό εγώ, ο οποίο δημιούργησε την δημόσια ιδιωτική εταιρική σχέση στα νοσοκομεία, στις δημόσιες, ε, στα δημόσια νοσοκομεία που πέρασαν σε ιδιωτική διαχείριση και ε, μπορέσαν έτσι να ε, μπορέσουν να στηθούν στα πόδια τους. Δεν μπορεί κανείς να μου κάνει μαθήματα σε σχέση με αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν πράγματα που μας οδηγούν σε μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Ευχαριστώ και τους δυο σας για τις παρατηρήσεις σας. Από πλευρά σα τώρα, εκπρόσωπε τη Επιτροπή, θα ήθελα να σα ζητήσω να τοποθετηθείτε για την έκθεση του κυρίου Μπουσόη και για άλλα θέματα που θα θέλατε να αναφέρετε για το πακέτο των εκθέσεών μα. Μετά θα λάβει τον λόγο ο κύριο Μπουσόη. Και μετά μία ή δύο ε, κατακλείδη παρατηρήσεις θα κάνω και αν η κυρία Κανιέται και ο κύριος ε, Κορέντε κάπως θέλουν να προσθέσουν κάτι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε στις 12.30 θα έλεγα. Η εκπρόσωπος τη Επιτροπής πρώτη παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μικροφωνίζει το τηλέφωνο. Ε, thank you, Chair. Συγγνώμη γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε έλεγα. Γενικά καλωσορίζουμε ευρύτερα το γεγονός ότι οι συγητές και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή προσπαθούν να εργαστούν στο να ταυτοποιηθούν προτεραιότητες και να εντοπιστούν προτεραιότητες. Αυτό καταδείχθηκε σήμερα και από τη συζήτηση. Είναι ένα δυσχερές εγχείρημα. Υπάρχουν πολλά θέματα που όλοι θα θέλαμε να αντιμετωπιστούν και που ειλικρινά 200 μέτρα ή δράσεις είχαμε όταν ξεκινήσαμε από πλευράς Επιτροπής σε αυτό το εγχείρημα. Όπως εσείς οι ίδιοι τονίζετε, υπάρχει ανάγκη να τεθούν προτεραιότητες για να είμαστε αποτελεσματικοί στο έργο μας. Ας θυμηθούμε ότι αυτό το οποίο στοχεύουμε να κάνουμε εδώ να πετύχουμε είναι μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρώπης. Τι θα μπορέσει να επιτευχθεί ως προτεραιότητα και με κατεπήγοντα χαρακτήρα. Σε αυτό επικεντρωνόμαστε τώρα όχι να ζητηθεί από την Επιτροπή να αναλάβει απλά μια νέα πρωτοβουλία, αλλά να συμφωνήσουμε ότι όλοι, όλοι ότι πρέπει να επιτευχθούν αυτά, να τα καταφέρουμε και γοργά κιόλα υπάρχει ένα στοιχείο εφικτού και βιωσιμότητα σε σχέση με αυτά τα μέτρα. Άλλα είναι πιο συγκεκριμένα, πιο εξειδικευμένα και πιο σωστά από άλλα. Η αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ε, προσόντων είναι υψηλά ως προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη. Εργαζόμαστε, εργαστήκαμε σκληρά γι' αυτό και από πλευράς ε, συναδέλφου που ε, είναι ε, έχει αρμοδιότητα για συζητήσεις με τους επαγγελματικούς κύκλους. Όλα αυτά δίνουν πρόσθετη αξία. Είναι εξειδικευμένα, αλλά όπως και προαναφέρθηκε από την κυρία Βάιλερ, πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή την πρόσθετη αξία και ότι θα λειτουργήσουν. Και δεν είναι δεδομένο ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να είναι βιώσιμα για όλους τους εμπλεκόμενους. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν με πολύ προσοχή για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Άλλα στοιχεία, δημόσιες συμβάσεις και αγορές. Εδώ αφορά αυτό πολλές πολιτικές και για την καινοτομία, για παράδειγμα, που θα συζητηθεί αυτό το απόγευμα εδώ από ό,τι με έχουν πληροφορήσει. Η κυρία Βάιλερ είπε ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει κατακαιρματισμός, κατάτμιση αυτής της ημερήσιας διάταξης από υπερβολικά πολλούς εμπλεκόμενους και μέτρα. Φυσικά θα πρέπει να ε, ε, επανορθώσουμε, να αντισταθμίσουμε όλα αυτά. Αλλά οι συμβάσεις, οι αγορές πρέπει να διαδραματίζουν το ρόλο τους υπό διαφορετικά πρίσματα και προσεγγίσεις. Το κοιτάζουμε, το εξετάζουμε πολυσχηδώς λοιπόν και σφαιρικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται και ε, από διάφορες πρωτοβουλίες που δείχνουν τα, τον εγκάρσιο χαρακτήρα, οριζόντιο χαρακτήρα και επιπτώσει αυτού του τομέα, επίσης καταδεικνύεται ότι έχει ένα μια πολύ μεγάλη ε, δύναμη αυτό το εργαλείο, μεγάλη δυναμικότητα. Θα θέσουμε την έμφαση στο να βρούμε τη σωστή ε, χρήση κονδυλίων από τους ε, πιο αρμόδιους ώστε να υπάρχει καλύτερη χρήση κονδυλίων διάθεση και χρήση τους. Και αυτό είναι ένα κύριο, κύριο θέμα για τις συμβάσεις και αγορές. Και ε, ολοκληρώνω. Ενθαρρύνεται ε, το έργο και οι προσπάθειες για τις ιδιωτικοποιήσεις, οι προσπάθειες ε, όλων των εμπλεκομένων και των εισηγητών. Πρέπει να χαιρετιστούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Και εγώ για το έργο που επιτελείτε στεναρά για αυτό το χαρτοφυλάκιο εσείς και που οι προσπάθειές σας είναι τόσο σημαντικές για μας. Εσείς κύριε Μπουσόη θα θέλατε να ανακεφαλαιώσετε υπό το πρίσμα σας. Ευχαριστώ θα μιλήσω ρουμανικά πρόεδρε για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ τον εισηγητή και Θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν εδώ για αυτή την έκθεση. Σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν. Και έτσι σίγουρα σε μια ιστερότερη χρονική στιγμή θα έχουμε ευκαιρία πιο διεξοδικά να τοποθετηθούμε για αυτό το θέμα και να ε, το συζητήσουμε ξανά. Προς την κυρία Γκέπχαντος αποδέκτη. Όταν κάνω λόγο για Silicon Valley στην Ευρώπη, το κάνω υπό το εξή πρίσμα. Έχοντας υπόψη συνολικά την υποστήριξη για την καινοτομία, δεν ήθελα η, απόλυτα να εκφανθώ, να, αποφασ... να τοποθετηθώ υπέρ του γαλλικού προτύπου όχι, πρόκειται εδώ για ομάδες ομαδοποιημένα και κατηγορίες επιχειρήσεων και για την προστασία του περιβάλλοντος πάντα, λαμβάνοντας υπόψη την αηφορία και τις πράσινες τεχνολογίες, προστασία περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, αηφορία στην ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι πτυχές που έχουν προτεραιότητα και ως προτεραιότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν. <clears throat> και εγώ είμαι με ανοιχτό πνεύμα αντιμετωπίζω οποιασδήποτε τροπολογίες που θα συνεισφέρουν σε βελτιώσεις σε αυτούς τους τομείς. Να προσθέσω κάτι άλλο. Προστασία περιβάλλοντος, όπως είπα, κλιματικές αλλαγές και αηφορία στην ανάπτυξη. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, να τοποθετηθώ για την επικοδομητική συνεργασία. Ήδη είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν με την κυρία Ρενιό και φυσικά αυτό που θα θέλαμε είναι να υπάρξει και ε, συμπερίληψη των ενεργειακών ε, πολιτικών για την ενέργεια και των πολιτικών για τις μεταφορές. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, για μια τροπολογία που ε, σκοπεύαμε να κατατεθεί, δεν υπήρχε όμως αρκετός χώρος για να ληφθούν υπόψη όλα αυτά και Φυσικά πρόκειται για θέματα, για ενεργειακά ζητήματα και για μεταφορές εδώ που αναφέρω. Τώρα για τις τοχυδρομικές υπηρεσίες δεν ε, σκεφτόμουν ε, την δημιουργία Ευρωπαϊκής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, παρότι θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα. Απλά ήθελα να υπάρξει σωστή υλοποίηση της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Φερρυπίν, μέτρα, υποστήριξη του ηλεκτρονικό ο τραπεζικός τομέας πρέπει να αναφερθεί βέβαια στην έκθεση. Περιμένω τροπολογία σχετικά. Τώρα για την, ε, την επαγγελματική ταυτότητα. Συμφωνώ ότι χρειάζεται να γίνει πρώτα μια μελέτη επιπτώσεων. Ξέρω ότι η Επιτροπή ασχολείται με το θέμα. Πριν από λίγο καιρό είχα συντάξει μια, ε, μάλλον ήμουν σκιώδη σε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Κάποιοι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν ότι αυτή η επαγγελματική ταυτότητα είναι χρήσιμη, άλλοι δεν τη θεωρούν και πολύ χρήσιμη γιατί πιστεύουν αποτελεί επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η ταυτότητα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Και θα μπορούσε να είναι μια πρόταση επιτροπής και αν κάποια επαγγέλματα θεωρήσουν ότι διευκολύνεται η κυκλοφορία των επαγγελματιών του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκολύνουν την αναζήτηση εργασίας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό. Επίσης, πιστεύω ότι η ενιαία θηρίδα είναι μια ιδέα που αξίζει να υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά το σημείο 18 να διευκρινίσω κάτι. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη αυτές τις αθέμητες εμπορικές ή, ή, εμπορικές πρακτικές που ε, επιβαρύνουν τους καταναλωτές Θέλω να εξετάσουμε επίσης και το πώς θα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις σχέσεις τους με τις μεγάλες. Δεν πρέπει ωστόσο να επηρεάσουμε την λειτουργία της αγοράς με τον τρόπο αυτό, απλά να φροντίσουμε ούτω ώστε να τηρούνται οι κανόνες. Να πω στην κυρία Ρούλη ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να έχει θέση στην έκθεση. Δεν είναι εύκολο τόσο να αποφύγουμε επικαλύψεις. Υπάρχουν ε, διαστάσεις που βρίσκονται και στις τρεις εκθέσεις. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο να έχουμε μια έκθεση συνεκτική και να μην επαναλαμβάνουμε τις ίδιες προτάσεις. Σε ό,τι αφορά τον οικολογικό φόρο. Είναι γνωστή πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να, διευκρινεί, να διευρύνουμε τα σημεία που αφορούν στην τυποποίηση. Ε, η τυποποίηση ήταν ένα σημαντικό ζήτημα στη συζητήση στην Επιτροπή και η τυποποίηση αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα καλό μέτρο ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. Έχω ένα σημείο που αναφέρεται στην τυποποίηση, θα μπορούσαμε να το δουλέψουμε περισσότερο. Τώρα για το ΦΠΑ το ερώτημα του κ. Κοσνούτσικ. Προφανώς δεν μπορούμε να μιλούμε για εναρμόνιση του συντελεστή ΦΠΑ στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, δεν θα πηγαίνω τόσο μακριά. Πιστεύω ότι μια, καλή, μια τέτοια πρόταση θα ήταν καλή. Το ίδιο αφορά και στην πρόταση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε ενιαία, ενιαίο συντελεστή στη φορολογική των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι ένα καλύτερο σύστημα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ διότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ κρατών μελών στην απόδοση του ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά τώρα την φορολογία των εταιριών, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του φάσματος της φορολογίας, όχι ε, ενιαίο συντελεστή. Η επιβολή του η, η επιβολή του φόρου είναι εθνική προτεραιότητα και μπορεί να ποικίλει από κράτο σε κράτο ή από περιφέρεια σε περιφέρεια. Θα σταματήσω εδώ γιατί ο κύριος Χάρμπορ μου κάνει σήματα ότι πρέπει να τελειώσω. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την υποστήριξή τη. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον κύριο Μπαρνιέ για το νομοθετικό αυτό κείμενο. Το single Market Act είναι εξαιρετικά καλό κείμενο. Πρέπει να περιοριστούμε στις βασικές μας προτεραιότητες. Όπως έλεγα, είχα υποβάλει μια τροπολογία για πέντε μέτρα προτεραιότητας, πέντε βασικά ζητήματα. Περιμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων, γιατί θα ήθελα να υιοθετήσω τις προτάσεις των συναδέλφων και να μην προχωρώ μόνο με τις δικές μου ιδέες. Περιμένω δε και την άποψη των διαφόρων επιτροπών για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Okay, well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ όλου. Νομίζω πως ήταν αξιόλογο το σημερινό πρωινό. Άξιζε να αφιερώσουμε το πρωινό στη συζήτηση αυτή τη σημαντικής έκθεσης και ήταν λογική και η απόφαση των συντονιστών να κάνουμε τρει εκθέσει γιατί είναι σαφέ πω έχουμε πολλέ πτυχέ να καλύψουμε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή αλλά και την Ουγγρική Προεδρία. Και ξέρω βέβαια πω οι ε, συνάδελφοι το παρακολουθούν πολύ στενά και θα θυμάστε πω και ο υπουργό, ε, όπω μα είπε την προηγούμενη εβδομάδα ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα και στις 31 ε, Μαΐου βεβαίως το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα εγκρίνει την τελική του θέση. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Η αρχική, τρο... η αρχική προθεσμία για τροπολογίες ήταν ε, στις 27 Φεβρουαρίου και μετά θα ψηφίσαμε στις 7 ε, Μαρτίου που θα ήταν στο Στρασβουργό. Είχαμε κάποιες προτάσεις ε, να έχουμε περισσότερο χρόνο για τροπολογίες χωρίς να μειωθεί ο χρόνος για να βρεθούν συμβαστικές τροπολογίες. Το εξετάσαμε αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν τροπολογίες μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, 5η, 12 η ώρα το μεσημέρι Οπότε θα έχουμε ολόκληρη τη βδομάδα του Στρασβούργου για να διαπραγματευτούν οι συγητές χωρίς ε, να μας εμποδίσει αυτό μετά να δούμε τις τροπολογίες 27 Φεβρουαρίου. Μου φαίνεται λογική αυτή η πρόταση. Οπότε αν συμφωνείτε με αυτό, τότε νομίζω να έχουμε 10 Φεβρουαρίου 12 ώρα το μεσημέρι ως προθεσμία για τις τροπολογίες. τελική προθεσμία, αν συμφωνούν και οι συγητές μας μετά 28 Φεβρουαρίου για να εξετάσουμε τις τροπολογίες και 7 Μαρτίου στο Στρασβούργο Δευτέρα για να ψηφίσουμε την πρόταση της ουσίας και θα έχουμε και όλες τις νομοδοτήσεις βεβαίως μέχρι τότε δεν θα αναφέρω τώρα όλους τους συγητές απλά να σας πω πως Έχουμε γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Απασχόλησης, Νομικών, Πολιτικών Ελευθεριών, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και ε, Αναφορών, τις οποίες ο Πρόεδρος θα μας πει κάποια πράγματα και ακούσαμε σήμερα ήδη από την Επιτροπή Μεταφορών, οπότε είναι ενδιαφέρον το ότι έχουμε τόσο πολλές επιτροπές που εμπλέκονται, αλλά είναι κάπως απογοητευτικό το ότι μόνο ο κ. Κρότσμαν είναι εδώ σήμερα από τους ΣΥΙΤΕΣ. Οπότε καλό θα είναι οι ΣΥΙΤΕΣ να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες επιτροπές. Ο κ. Μπουσόη νομίζω ήθελε να επανέλθει. Ναι, ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το λύσουμε. Στις 28 είναι ομάδα των ομάδων και η ομάδα μας θα είναι στην Κοπενχάγη. Οι φιλελεύθεροι θα λείπουν δηλαδή επισήμως από τις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο θα είναι πρόβλημα για μένα αλλά εάν δεν υπάρχει άλλη λύση μπορεί ίσως η συζήτηση και η ψηφοφορία να γίνουν μαζί. Μπορούμε να τα στείλουμε και με email βεβαίως στη γραμματεία, απλά να ξέρετε το πρόβλημα αυτό που έχουν οι φιλελεύθεροι. Το πρόβλημα, Κρίστιαν, είναι πως 28 Φεβρουαρίου είναι η μόνη ημερομηνία που υπάρχει μέχρι από τώρα μέχρι την ψηφοφορία και υπάρχει μόνο μια μισή ώρα που έχουμε στο Στρασβούργο, οπότε δεν μπορούμε να εξετάσουμε, δεν έχουμε χρόνο να εξετάσουμε τι τροπολογίε. Βεβαίω μπορεί να τα υποβάλει γραπτό ή να ορίσεις κάποιον από την ομάδα σου να κάνει σχόλια για το που βρισκόμαστε. Καταφέραμε λοιπόν να βρούμε ένα συμβασμό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Αυτό ήταν ο καλύτερο. Οπότε σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω τρει η ώρα ακριβώς να είστε εδώ γιατί θα είναι εδώ η Επίτροπο, η Γκάγκεν Κουίν να μιλήσει για την καινοτομία και τις δημόσιες προμήθειες. Παρακαλώ λοιπόν τρεις η ώρα